Ξεκινάμε συνάδελφοι. Ζητώ συγγνώμη για την ε, δεκάλεπτη καθυστέρηση. Πάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά η οργάνωση της επίσκεψης στο Βερολίνο. Επίσης, μίλησαν για, την, για τον καθορισμό του προγράμματος ε, στη Ρουμανία. Του ζήτησαν να το κάνουν το συντομότερο δυνατόν οι συνάδελφοι που εκπροσωπούν την κάθε ομάδα. Για τις αποστολές του 2012 λάβαμε από την Προεδρία το χρονοδιάγραμμα. Άκουσα διάφορες φήμες για την προηγούμενη απόφαση που ελήφθη. Προσπαθούν να υποσκάψουν την αξιοπιστία της πλειοψηφίας μας. Είναι σκάνδαλο. Και ελπίζω να μην συζητηθεί και να μην αμφισβητηθεί. Για το χρονοδιάγραμμα των αποστολών του 2012, η ομάδα των συντονιστών απάντησε στο, στο Προεδρείο, το οποίο ζήτησε περισσότερες λεπτομέρειες για όσους θα συμμετάσχουν στις αποστολές και για τους προορισμούς. Επιβεβαιώσαμε κάποιες χώρες που θέλουμε να επισκεφτούμε πέρυσι, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Γαλλία και, και προσθέσαμε και τους δύο προορισμούς που στις προηγούμενες συνεδριάσεις ε, το συντονιστό είχαν αναφερθεί, Ισπανία και Γερμανία. Το λεπτομερές πρόγραμμα θα καθοριστεί, θα καθορίζεται κάθε φορά. Αν, ανεπίσκεψη δηλαδή. Οι συντονιστές αποφάσισαν ε, και για τον ε, συντάκτη της γνωμοδότησης για το έτος ε, του Ευρωπαίου πολίτη του που είναι το 2013 από την ομάδα EFD. Επίσης, Επίσης, ο πρόεδρος της Επιτροπής ΑΦΚΟ μας έκανε μια ανακοίνωση για τον τρόπο με τον οποίο θα συλλέξουμε πληροφορίες για τη λαϊκή πρωτοβουλία. Θα συλλέξουμε, συγγνώμη, υπογραφές για τη λαϊκή πρωτοβουλία και ζήτησαν από την Επιτροπή μας να συντάξουμε μια γνωμοδότηση μέχρι αύριο για το θέμα αυτό. Όπως είπα χθες, στη συνεδρίασή μας το Κοινοβούλιο έλαβε μια καταδικαστική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την περίπτωση Τέγκε Μπάουερ, που είναι μια αναφερόμενη, που επειδή ε, απορρίψαμε την αναφορά της εδώ στην Επιτροπή το 2007, ε, επειδή δεν ήταν παραδεχτή έκανε προσφυγή. Το δικαστήριο θεωρεί ότι η Επιτροπή μας πρέπει κάθε φορά να δικαιολογεί την δήλωση του παραδεκτού ή του μη παραδεκτού. Και οι συντονιστές σημείωσαν αυτή τη διαδικασία, ότι ξεκινάει δηλαδή αυτή η διαδικασία, αλλάζει ο τρόπος που συντάσσουμε τις, αποστο... τις επιστολές, ε, ειδικά για αναφορές που θεωρούνται μη παραδεκτές. Σε ό,τι αφορά την ε, συνεδρία που θα κάνουμε στις 21 και 22 Νοεμβρίου, Έχουμε ένα σχέδιο ημερήσια διάταξη το οποίο θα μοιραστεί τις επόμενες ώρες, ούτω ώστε να εγκριθεί, γιατί χθε δεν ήταν έτοιμη αυτή η ημερήσια διάταξη. Αυτά αποφάσισαν οι συντονιστέ. Κλείνουμε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη και πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξη. διάταξης. Το σημείο 14 δηλαδή, Έχουμε την εισηγήτρια την κυρία Βαλεάν, έκθεση του 2010 για την Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα χαιρετίζοντα όλες τις προσπάθειες που έκανε η Επιτροπή μέχρι τώρα προκειμένου να ενισχύσει την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας γιατί αυτός είναι και ο στόχος της έκθεσης αυτής που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2010. Συζητώντα την έκθεση αυτή τώρα για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, πρέπει να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι το σώμα πολλές φορές μέχρι τώρα έχει υπογραμμίσει τη σημασία που έχει να είναι πιο αποτελεσματική και πιο εύκολη χρήση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Το έχουμε υπενθυμίσει πολλές φορές αυτό. Έχουμε έκθεση όσον αφορά την ε, εφαρμογή της οδηγίας 38 για την μετακίνηση των μελών των ε, οικογενειών ε, πολίτη κράτους μέλους και έχουμε αναφέρει τα εμπόδια που υπάρχουν όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία για τη μετακίνηση λοιπόν ε, ατόμων που δεν είναι μέλη της, από μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όμως αποτελούν μέλη οικογένειας ατόμου που είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολη η εγκατάστασή τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε επίσης μια έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, είτε από το 2008, όπου υπογράφονται τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Η έκθεση πολύ καλά περιγράφει διοικητικές δυσκολίες και καταλήγει στο ότι η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να χτίζεται γύρω από τα δικαιώματα και τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών και να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Επίσης είχαμε και άλλη έκθεση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τις προπτικές με το θέμα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και αυτό έγινε το 2009 εξακολουθούν, διαπιστώνουμε στην έκθεση αυτή, να υπάρχουν εμπόδια για την επανένωση οικογενειών και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει κατάλογο με όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Έπειτα, το θέμα του προγράμματος εργασίας όσον αφορά την δικαιοσύνη και ελευθερία για την περίοδο μέχρι το 2014 βάζει τον Ευρωπαίο πολίτη στην καρδιά των ευρωπαϊκών πολιτικών. Είμαι συγκίτρια λοιπόν για την έκθεση αυτή του 2010 όσον αφορά την άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα έλεγα να επικεντρωθούμε στις δράσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή ε, βάσει των αναφορών που έχουν φτάσει στην Επιτροπή μας κατά την περίοδο 2008-2010. Για το σκοπό αυτό πάνω από 300 σχετικές αναφορές εξετάστηκαν από εμάς. Δεν μπορούμε βέβαια στην έκθεση αυτή να εξετάσουμε όλα τα εμπόδια που εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που είναι 25 κύρια εμπόδια. Εγώ προτείνω να επικεντρωθούμε σε μερικά προβλήματα τα οποία αναφέρονται πολύ συχνά στις αναφορές που φτάνουν στην Επιτροπή μας. Κυρίως πρόκειται για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, Πρόκειται για την κοινωνική ασφάλιση και για την μη αναγνώριση των ε, τίτλων σπουδών ή προσόντων. Έχω ήδη μοιράσει μια, ένα επεξηγηματικό σημείωμα όσον αφορά τα εμπόδια αυτά και δεν θα σας τα επεξηγήσω τώρα όλα, εκτός αν μου το ζητήσετε. Μερικά πραγματάκια. Πρώτα για την ελεύθερη κυκλοφορία. Όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει το δικαίωμα αυτό για τους πολίτες μας. Είναι ένα πολύ γνωστό δικαίωμα. 88% των Ευρωπαίων ερωτηθέντων αναγνωρίζουν αυτό το δικαίωμα. Όμως, όμως Το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, παρόλο που αναγνωρίζεται ευρέως από τους Ευρωπαίους πολίτες, εξακολουθεί να είναι εκείνο το οποίο έχει αναπτυχθεί λιγότερο από τις τέσσερις ελευθερίες που αναφέρονται στη συνθήκη. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία. Έρχομαι τώρα στο θέμα της κοινωνικής ε, ασφάλειας. Είναι βέβαια περίπλοκη η νομοθεσία και δύσκολα την κατανοούν πολλές φορές οι πολίτες και από την άλλη μεριά οι αρμόδιες αρχές δεν εφαρμόζουν πάντα σωστά τα όσα προβλέπονται για την κοινωνική ασφάλιση. Τέλος, για την αναγνώριση τίτλων σπουδών ή προσόντων, εδώ θέλουμε φυσικά να εφαρμόζεται η Οδηγία 36 του 2005. Αλλά ε, ενίοτε είναι ανεπαρκής η μεταφορά της στην Εθνική Νομοθεσία. Τίθεται θέματα υπηκότητας για ορισμένες χώρες μέλη. Και πριν τελειώσω την σύνοψη αυτή της εκθεσής μου, θα έλεγα, όπως είπε και ένας συνάδελφος, ο κύριος Λόου, μάλλον από τη γραμματεία το έλεγε, ότι πολύ σημαντικό στην έκθεση είναι να υπογραμμίσουμε, να τονίσουμε το δικαίωμα στις αναφορές που έχουν οι πολίτες μας. Έτσι διευκολύνεται και το δικό μας το έργο και έχουμε την ευκαιρία να προβληματιστούμε για το πώς ε, ε, δουλεύουν οι ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένω σχόλια από τους συναδέρφους και εφόσον μπορώ θα ήθελα να ξαναπάρω το λόγο στο τέλος για να σας αναφέρω και το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Βαλεάν για τη δουλειά σας και για την παρουσίαση που μας κάνατε. Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, η κυρία Γεωργιάδου έχει το λόγο παρακαλώ. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Να πω καταρχήν ότι χαιρετίζουμε ε, πολύ θετικά την επικείμενη έκθεση. Η... Πέρα από τις 25 δράσεις ε, για την έκθεση για τους πολίτες, σκοπός ήταν να ανοίξει συζήτηση και με το Κοινοβούλιο, με άλλα θεσμικά όργανα, με όλους τους βασικούς εμπλεκομένους Προτείναμε επίσης να ορίσουμε το 2013 το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών ώστε να ε, αποκτήσουν ορατότητα τα θέματα της ηθαγένειας και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις εκλογές επίσης το 2014, συμμετοχή στις εκλογές, εκλέγην κλπ. Οπότε θεωρήσαμε ότι θα ήταν ευκαιρία να προχωρήσουμε το θέμα αυτό, αυτή η περίοδος και έτσι θα μπορούσαμε να δούμε πώς θα ε, καταρρύπταμε όλα αυτά τα εμπόδια για τα, στα δικαιώματα των πολιτών. Η Επιτροπή σας είναι από τις πιο σημαντικές διάβλους επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των ε, θεσμικών οργάνων της Ένωσης, άρα είναι και στο προσκήνιο η Επιτροπή αυτή όταν πρόκειται να εισακουστούν τα μελήματα, οι προσδοκίες των πολιτών και να εντοπιστούν κενά και ε, επίμονα προβλήματα. Οπότε προσβλέπουμε με ενδιαφέρον στη στενή συνεργασία μας μαζί σας για να συνεχιστεί η διαδικασία αυτή με τρόπο θετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπρέντεν Γκάστ, ξέρω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με την, ε, τα δικαστικά προβλήματα, επιμέλεια κλπ. Πολλές φορές είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουν οι γονείς προβλήματα, διότι είναι πολύ περιοριστική η όρη για την επιμέλεια. Ε, στα παιδιά είναι σημαντικό αυτό. Εγώ στο και είχα εμπειρία από τη, τις διαδικασίες διαζυγίων και πήρα πολλά αιτήματα από γονείς εκ των οποίων ο ένας πηγαίνει να εγκατασταθεί σε άλλη χώρα, προβλήματα με τα παιδιά, ε, τα νόμιμα δικαιώματα των γονέων, δικαιώματα επισκέψεων κλπ. Ε, τα προβλήματα είναι πολλά γιατί είναι και πολλά τα προβλήματα και οικονομικά και γλωσσικά κλπ. Δεν ασχολείται με τα θέματα της επιμέλειας των τέκνων άμεσα το δίκαιο της Ένωσης, αλλά Όλες οι χώρες της Ένωσης αναγνωρίζουν το δικαίωμα άμεσης επαφής και σχέσεων και με τους δύο γονείς για το συμφέρον του παιδιού. Επίσης όλες τις χώρες με την εξαίρεση της Δανίας το πιο κοντινό δικαστήριο της συνήθους διαμονής επιλαμβάνεται την εκδίκαση θεμάτων γονεϊκής ευθύνης. Δυστυχώς υπάρχουν δυσκολίες στο πώς ερμηνεύεται η συνήθις διαμονή. Το η νομολογία του δικαστηρίου εξεδίκασε ε, μια υπόθεση, είναι 23 του 07, αλλά ε, ως επιτοπλίστων ε, ε, ορίζεται η υπόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2009. Δεν υπάρχει λοιπόν εναρμονισμένη ερμηνεία. Επίσης το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει ότι οι αποφάσεις σχετικά με την επιμέλεια αναγνωρίζονται αυτομάτως και εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε το πρόβλημα ως το μεγαλύτερο πρόβλημα ως το πρόβλημα της πρόσβασης στο δικαστήριο το οποίο θα αποφασίσει με το καλύτερο ε, συμφέρον του παιδιού κατά νουν, ε, με βάση ε, κατάλληλης παροχής πληροφοριών. Αυτό ισχύει για όλους τους πολίτες της Ένωσης ανεξάρτητα από την ηθαγένειά τους. Κυρία Ζανόγκα, ευχαριστώ. ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Βαλεανό, την εισηγήτρια, η οποία μας έδωσε πολύ περιεκτικά στοιχεία για την πρώτη μας συζήτηση και ελπίζω στην περαιτέρω συνεργασία μας. Πόσο μάλλον που Είμαι σκιώδης από τους πράσινους σε αυτή την ε, έκθεση των Κομισιών και επίσης και για την έκθεση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για το ίδιο θέμα. Να υπογραμμίσω καταρχήν ότι όλα τα προβλήματα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό για τη συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντικά το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία πρώτα απ' όλα και υπάρχουν και πολλές αναφορές ε, πάνω σε αυτό το θέμα. Επίσης, ε, θέματα κοινωνικής ασφάλισης, αναγνώρισης διπλωμάτων, προσόντων και πολλά κοινωνικά θέματα επίσης. Τώρα, για το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεσθε, στις ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές παρά το γεγονός ότι το 2010 δεν ελάβαμε και τόσες πολλές αναφορές για αυτό το θέμα. Παρόλα αυτά πρέπει να αναφέρουμε τα προβλήματα Υπήρχε μια περίπτωση λέει, από τη Λετωνία με 16.000 υπογραφές για το δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές και δημοτικές εκλογές. Το αίτημα εξετάστηκε το 2008 και συμπεριελήφθη στην έκθεση της Επιτροπής Αναφορών. Έγινε παραδεκτή το, την άνοιξη του 2009 και να αναφέρουμε και μια άλλη αναφορά από την Εσθονία πάλι συλλογική αναφορά, την εξετάσαμε το Φεβρουάριο τρέχοντος έτους και αφορά το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές της ευρωπαϊκές Το θέμα της ε, μόνιμης ε, παραμονής είναι θέμα γιατί το 20% των Λετωνών έχουν πρόβλημα γιατί κάποιοι είναι ανιθαγενείς και κάποιοι άλλοι είναι, ε, έχουν την ηθαγένεια συνήθως γειτονικών χωρών, της Ρωσίας ως επιτοπλίστων. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγην στις δημοτικές εκλογές, δεν έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγεσθε. Ούτε ε, μπορούν να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές εκλογές. Τώρα, για τους Λετωνούς, ε, ε, και αυτοί είναι 20%, ή μάλλον τους μη Λετωνούς, οι περισσότεροι όμως είναι ανηθαγένεις. Έχουν ειδικό καθεστώς που τους επιτρέπει να επιστρέφουν στη Λετωνία και να προστατεύονται από, τις, από το λετωνικό κράτος όταν είναι στο εξωτερικό, αλλά οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούν να μην έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκλογές. Δεν έχουν δικαίωμα ούτε του εκλέγην ούτε του εκλέγεστε. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε πεδίο εργασίας μεγάλο, με βάση τις αναφορές που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Αναφορών, ώστε να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Με βάση, είπαμε, την έκθεση που ελάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και, αν μου επιτρέπετε, να προσθέσω ότι Υπάρχουν και πιο θεωρητικά και πολιτικά ζητήματα που αναφέρονται στην ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέματα τα οποία δεν έχουν ε, καταλήξει σε συνένεση από τα ε, ευρωπαϊκά κόμματα, ενώ είναι θέματα προστιθέμενης αξίας για την ηθαγένεια της Ένωσης. Ποια είναι, υπάρχουν διαφορές μεταξύ εθνικής ηθαγένειας και ενωσιακής, αν θέλετε, ηθαγένειας. Κατά την προηγούμενη θητεία μας ε, είχαμε μια έκθεση που ετοιμάστηκε από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Από, ε, την, ε, η έκθεση Κατάνη από, τη, από βουλευτή της Αριστεράς με επαναστατικές προτάσεις μεταξύ άλλων για τη νέα ηθαγένεια, η οποία δεν θα είναι υποχρεωτική, θα απορρέει από την εθνική ηθαγένεια και θα χορηγείται όταν υπάρχει, ας πούμε, ε, περίπτωση ανιθαγενών με μόνιμη παραμονή ή από, σε ε, ανθρώπους με ηθαγένεια τρίτων χωρών. Δεν πέρασε όμως από την Ολομέλεια η πρόταση αυτή. Όμως, παρόλα αυτά, μπορούμε να φρεσκάρουμε λίγο τη συζήτησή μας επί των ε, απόψεων αυτών, με αυτή την ευκαιρία τώρα. Η πρότασή μου σχετικά με την ε, έκθεση είναι να αναφέρομαι τις ε, προτάσεις αυτές τις παλιότερες, γιατί εξακολουθούν να υφίστανται σε ευρύτερους ε, ε, κύκλους, αν θέλετε, των πολιτών μας. Ελπίζω λοιπόν ότι θα γίνει καλή η έκθεση αυτή και θα φέρει νέες ιδέες για να βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτά όλα τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σκιώδης συγγήτρια κάποια ομάδας. Ε, αν κάποιος προηγείται, ας πάρει το λόγο πριν από μένα. Είναι νωρίς ακόμα, δεν έχω ξυπνήσει. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής. Ως μέλος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ παίρνω το λόγο και είμαι ευρωβουλευτής που έχει μεγάλη δράση στον τομέα αυτό. Μ' αρέσει το γεγονός ότι ασχολείστε με αυτή την έκθεση στην Επιτροπή σας και συγχαίρω την κυρία Βαλεάν που εντόπισε, εστίασε τα βασικά προβλήματα που έχουμε. Αυτό που με εκπλήσει είναι ότι κάνουμε κύκλους σε αυτό το θέμα, πραγματικά, σας το λέω ειλικρινά. Η οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία έχει παλιώσει, έχει 7 χρόνια στην πλάτη και τέθηκε σε ισχύ πριν από 5 χρόνια. Και ακόμα, παρόλα αυτά, έχουμε μεγάλα προβλήματα για τους πολίτες και κυρίως με τα μέλη της οικογένειας ε, ατόμων από τρίτες χώρες. Δεν αναγνωρίζονται τα δικαιώματά τους. Βασικά είναι τρία τα μεγάλα προβλήματα. Αυτά μου λένε. Το πρώτο αφορά τις άδειες διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη χώρα μου δηλαδή, και ξέρω ότι αυτό υπάρχει και στην έκθεση της Επιτροπής σας πέρυσι, καθώς και στην γνωμοδότηση της Αιγύτριας, το θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Και θα ήθελα να το ψάξουμε λίγο περισσότερο, να το σχολιάσω. Θα ήθελα δηλαδή να δω τι πέτυχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθυνόμενη στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατά πόσο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει βελτιώσει τις διοικητικές πρακτικές του. Έχω αλληλογραφία για καθυστερήσεις, για κρατήσεις διαβατηρίων, διαβατήρια που δεν επιστρέφονται δηλαδή κτλ. κτλ. Ίσως θα το ψάξω διμερώς με την Κομισιόν να δω τι έχει γίνει. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν είμαστε χώρα Σέγγεν και τα μέλη της οικογένειας των Βρετανών πολιτών ή το νομίμος διαμενόντων. Ας τους αφήσω αυτούς έξω. Κυρίως τα μέλη της οικογένειας των ε, Βρετανών πολιτών που θέλουν ε, θεωρήσεις Σέγγεν και τουριστικές θεωρήσεις ακόμα. Αλλά κυρίως ε, δικαιώματα διαμονής ε, σε ένα άλλο κράτος μέλος. Αυτό είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και αρνήσεις χορήγησης των θεωρήσεων. Δεν υπάρχει σαφήνεια για τη διαφορά ε, για την ε, πληρωμή όχι της ε, θεώρησης αυτής καθεαυτής, αλλά για την πληρωμή ενός τέλους, γιατί η διαδικασία διεκπεραιώνεται από εξωτερικές υπηρεσίες. Το τρίτο πρόβλημα που θα το συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα είναι τα ζευγάρια ίδιου φίλου, ε, τα οποία είναι είτε παντρεμένα, είτε έχουν, ε, βρίσκονται σε ένα καθεστώς ε, επίσημο συμβίωσης. Έχουν θέματα δικαιωμάτων, θέματα αναγνώρισης του καθεστώτος, το κατά πόσο αναγνωρίζονται τα δικαιώματα κληρονομιάς τους. Ξέρω ότι υπάρχουν τέτοιες αναφορές ειδικά για αυτό το θέμα και θα επανέλθω σήμερα το απόγευμα σε αυτό. Αλλά πραγματικά έχω μπερδευτεί, γιατί τα είχαμε συζητήσει αυτά με την Αντιπρόεδρο Ρέντιγκ πέρυσι το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο. Του στείλαμε επιστολή και η απάντηση της με εκπλήσει. Είπε ότι οι πολίτες της Ένωσης που λείβουν που ζουν στα πλαίσια ενό γάμου ή μια σχέση αναγνωρισμένη θα πρέπει να κρατούν το καθεστώ αυτό και τα δικαιώματά του όταν μετακινούνται από ένα κράτο σε ένα άλλο. Θα έπρεπε. Αλλά δεν τα έχουν αυτά τα δικαιώματα. Γιατί δεν υπάρχει απόλυτο δικαίωμα με βάση την οδηγία του 2004. Υπάρχει μια κάποια, θα έλεγα παρόλα αυτά, διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους προορισμού. Να μην αναγνωρίσει, παραδείγματος χάρη, αυτή την ε, επίσημη συμβίωση. Ε, και δεν θεωρεί ότι είναι ότι συνάδει με το καθεστώς που προβλέπει για τα παντρεμένα ζευγάρια εκεί. Θέλω η Κομισιό να μου πει αν κάνει κάποιες διαδικασίες ε, επί παραβάση εναντίον κάποιων κρατών μελών. Έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες. Από την αλληλογραφία που είχαμε την κυρία Ρέντινγκ, γίνεται λόγο, για την απάντησή μας μιλάει για, μιλάει για διάλογο με τα 27 κράτη-μέλη. Ε, στην έκθεση του φθινοπόρου του 2010 γίνεται λόγος για αυστηρή εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κομισιόν ε, λαμβάνει μέτρο τόσο ώστε να εφαρμοστούν πλήρως οι διατάξεις της οδηγίας για την ελεύθερη α, κυκλοφορία. Αυτό τι σημαίνει, δεν σημαίνει και διαδικασίε επί παραβάση. Πότε θα ακούσουμε κάτι δημόσιο, πότε θα στυλιτεύεται ένα κρατό μέλο. Γιατί αυτή είναι μια εμβληματική πολιτική. Είναι κάτι που οι πολίτε μα, και ακόμα και οι δικοί μου πολίτε, οι Βρετανοί πολίτε που, είναι και τόσο, που δεν λατρεύουν τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεωρούν αυτά δεδομένα. Δεν καταλαβαίνουν μερικέ φορέ βέβαια ότι είναι χάρη στο ενωσιακό δίκαιο, ε, λένε Α, εντάξει θα πάω στην άλλη χώρα, εκεί θα, εκεί θα σπουδάσω, θα πάω να περάσω τη σύνταξή μου σε μία άλλη χώρα, σε μία τρίτη χώρα και νομίζω ότι όλα αυτά έτσι εμφανίζονται εν κενό, ξαφνικά, εν μία νυχτή. Δεν καταλαβαίνω που προέρχονται. Παρ' όλα αυτά τα εκτιμούν, τα θέλουν. Και είναι κρίμα και ντροπή και δεδομένου του εθροσκεπτικισμού που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κρίμα λοιπόν έλεγα ε, που δεν καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα. Το τελευταίο θέμα είναι. Το τελευταίο θέμα που θέλω να αφήξω. Ε, τα έχουμε μπερδέψει. Ποιος λύνει ποιο πρόβλημα, ποιο site ε, είναι υπεύθυνο, ποιο δίκτυο, έχουμε το Solvit, έχουμε ένα κάρο δίκτυα. Όλα αυτά με μπερδεύουν. Έχουμε τελικά μία πύλη προς την οποία απευθυνόμαστε. Υπάρχει μία ένας αποδέκτης για να λαμβάνει όλα τα προβλήματα και να τα επιλύει. Και αν δεν υπάρχει, πότε θα δημιουργηθεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουλάν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για την εισηγήτρια, για τους συναδέλφους, εγώ είμαι σκιώδης εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ την κυρία Βαλεάν για το εγγραφό της που μας έδωσε πολύ καλά συνοψίζει τι διάφορε ελλείψει του συστήματο μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων ελεύθερη κυκλοφορία, κοινωνική ασφάλιση και αναγνώριση τίτλων και προσόντων, όπω το δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε κλπ. Επίσης, χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι αναφέρεστε και στο δίκαιο τη οικογένεια και την... Ε, ε, ποιος αναλαμβάνει τα παιδιά σε περίπτωση διαζυγίου είναι πολύ καλό και εμείς ε, είχαμε πει ότι θέλουμε όλο και περισσότερο να λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις αναφορές που μας έρχονται για αυτά τα θέματα. Και θα πάμε και στο Βερολίνο μάλιστα για να εξετάσουμε ένα τέτοιο θέμα. Η έκθεση αυτή λοιπόν αναφέρεται σε πολλά ζητήματα και άρα μπορεί να υπάρξουν πολλές και διαφορετικές προβληματικές. Το δικαίωμα ε, αναφοράς των Ευρωπαίων πολιτών, για παράδειγμα, το θέμα της απασχόλησης, της δημιουργίας επιχειρήσεων, το θέμα της εθελοντικής εργασίας, ε, τράπεζες κλπ. κλπ, κλπ. Πάρα πολλά θέματα. Η ηθαγένεια είναι ένα θέμα που δημιουργεί μεγάλη αίσθηση πρέπει να έχουμε παραδείγματα από αναφορές για να καταδεικνύουμε τι ζητούν ε, οι πολίτες και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν όσον αφορά τα δικαιώματά τους. Αλλά όχι μόνο. Το θέμα της ηθαγένειας είναι ε, να αποφασίσουμε το εξή. Έχουν δικαιώματα οι πολίτες, συγχρόνως όμως έχουν και ε, υποχρεώσεις. Το ένα δεν πάει χωρίς το άλλο και πολύ συχνά ε, διαπιστώνουμε ότι οι πολίτε ενδιαφέρονται για την Ευρώπη όταν κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να έχουμε μια έκθεση που να αναφέρει και τα θετικά από την ηθαγένεια. Δεν έχει νόημα να επεκτηνόμαστε υπερβολικά πάνω στι έννοιε. Πρέπει να είμαστε πιο πρακτικοί και να χρησιμοποιούμε παραδείγματα συγκεκριμένων αναφορών, όπω έχετε κάνει κι εσεί, ε, ε, κυρία Συγγήτρια, στην έκθεσή σα. Γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε καλύτερα ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ευρωπαίο πολίτη είτε ως ιδιώτης, είτε ως καταναλωτής, είτε ως οικονομικός παράγοντας όταν παρεμβαίνει με μία αναφορά. Για παράδειγμα, η ελευθερία κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια είπατε ότι είναι το πιο δημοφιλές δικαίωμα. Αλλά είναι και η ελευθερία που έχει αναπτυχθεί περισσότερο. Τι δείχνει αυτό, ότι δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση. Ο Ζωφρασού για παράδειγμα, ένας ακαδημαϊκός Γάλλος, έλεγε ότι ο δημοκρατικός πολιτισμός βασίζεται στην ακρίβεια της ενημέρωσης. Εάν ο πολίτης δεν είναι καλά ενημερωμένος, τότε δεν σημαίνει τίποτα το να πηγαίνει και να ψηφίζει. Άρα λοιπόν για να δώσουμε ένα νόημα στις ευρωπαϊκές εκλογές πρέπει να ενημερώνουμε τον πολίτη, να πληροφορείται, να φτάνει και τελευταία πληροφορία μέχρι σε αυτόν. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει το δυνατό σημείο της έκθεσής σας, συνδυασμένο με το έτος 2013 που είναι ενημέρωση του πολίτη και πριν περάσουμε στην ε, εφαρμογή της πρωτοβουλίας των πολιτών. Τέλος, θέλω εκ μέρους του ΕΛΚ να σας πω ότι θέλω να συνεισφέρω σε συνένεση, χωρίς όμως να αφήσουμε απ' έξω οποιοδήποτε θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ερώτηση που απευθύνεται προς την Κομισιόν. Θέλει να απαντήσει η Κομισιόν τώρα. Μπορεί. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Θέλω να επικεντρωθώ στα μέτρα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ακολουθεί μια αυστηρή πολιτική όσον αφορά την εφαρμογή που αποτελείται και από διάλογο και από διαδικασίες επί και χαιρόμαστε που είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε ότι φέτος οι περισσότερες χώρες μέλη τροποποίησαν ή βρίσκονται στη διαδικασία τροποποίησης της νομοθεσίας τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν ε, προβλήματα και αδυναμίες που εντοπίστηκαν και συζητήθηκαν μαζί τους στο πλαίσιο του διαλόγου που έχουμε με αυτές τις χώρες. Στείλαμε και κοινοποιήσει σε 10 χώρες μέλη επίσημα και τώρα είμαστε στην διαδικασία ανάλυσης των απαντήσεων όσων έχουν ήδη απαντήσει. Σας διαβεβαιώνω δηλαδή ότι η διαδικασία αυτή είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται και που παρακολουθούμε στενά την νομοθεσία και τις πρακτικές που ακολουθούν οι χώρες μέλη. Όσον αφορά τώρα το ειδικό θέμα που αναφέρατε για το Ηνωμένο Βασίλειο με τις μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά την επεξεργασία και τις ε, διαδικασίες είχαμε διάλογο με τις Βρετανικές Αρχές που κατέληξε σε ένα σχέδιο από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, για παράδειγμα αύξηση του αριθμού περιπτώσεων που επεξεργάζεται. Υπήρχε μια αύξηση 400% ή να υπάρξει μια τηλεφωνική γραμμή ή γραμμή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου να υποβάλλονται τα διάφορα έγγραφα. Το Ενωμένο Βασίλειο δηλαδή κοινοποίησαν τον Οκτώβριο του 2010 σε εμά ότι ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό του φόρτου των αιτήσεων και ότι είναι μέσα στην προθεσμία έτσι όπως προβλέπεται από το κοινοτικό νόμο. Το Φεβρουάριο στείλαμε επιστολές σε πολίτες οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν σε εμά, τους ενημερώσαμε για αυτές τις εξελίξεις και τους ζητήσαμε να μας πούν μέσα σε τέσσερις εβδομάδες κατά πόσο πρόκειται για παράβαση όχι. Τέτοιες πληροφορίες ε, δεν πήραμε που να λένε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Εμεί όμω παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι συμμορφώνονται οι αρχέ με τι προθεσμίε όπω προβλέπονται στην οδηγία και θα επεξεργαστούμε κάθε νέο πρόβλημα ή αδυναμία που θα προκύψει ανάλογα με την κατάσταση. Η κυρία Βάλιαν τώρα για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ συνάδελφοι για τα όσα είπατε. Φυσικά και θα κάνω ό,τι μπορώ για να συμπεριλάβω τα σχόλιά σας στην έκθεσή μου. Μα υπάρχουν τόσα πολλά θέματα. Δεν υπάρχει μόνο η έκθεσή μου, υπάρχουν και ένα σωρό θέματα τα οποία προκύπτουν και τα βλέπουμε και στην τηλεόραση. Λοιπόν, για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών πρώτα απ' όλα. Φυσικά και υπάρχουν ακόμα εμπόδια και ένα σωρό θέματα που προκύπτουν όσον αφορά τους πολίτες τρίτων χωρών. Αλλά έχουμε και ένα σωρό θέματα που έχουν να κάνουν με Ευρωπαίους πολίτες. Δυστυχώς υπάρχουν δεκάδες μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες καταγγέλνουν θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος, που άπτονται των δικαιωμάτων. Δεν έχουμε βέβαια αναφορές για τους Ρώμα. Υπάρχουν δηλαδή και ένα σωρό άλλα θέματα τα οποία δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προτείνουμε λύσεις. Χρονοδιάγραμμα τώρα για την έκθεσή μου. Θα εξεταστεί στη, η έκθεσή μου στην Επιτροπή μας στις 20 Νοεμβρίου. Τέλη Νοεμβρίου, 29 Νοεμβρίου δηλαδή, είναι η προθεσμή για κατάθεση τροπολογιών. Ελπίζω να εγκριθεί η τελική μου έκθεση την συνεδρίασή μας του Ιανουαρίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα λίγο πολύ. Από εδώ και πέρα περιμένω τροπολογίες από εσά προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το κείμενό μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Βαλιάν. Έχουμε χρόνο λοιπόν για να συμπεριλάβουμε και τα σχόλια που ακούσαμε σήμερα από τους συναδέλφους, ούτως ώστε να φτάσουμε ε, προετοιμασμένη στην ε, Ολομέλεια. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Πάμε στο σημείο 15 δηλαδή. Έχουμε την αφορά 622 του 2010 και την 628 του 2011. Ένας από τους αναφέροντες είναι παρόν. Όχι και οι δύο, διορθώνει πρόεδρος. κύριος Γκάμπριελ Βοητσουλέσκου έχει το λόγο. Πρώτος. Ευχαριστώ τους Ευρωβουλευτές για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε την ε, ε, αναφορά μας για το σημείο αυτό και ευχαριστώ και την Επιτροπή για την ε, απάντησή της. Είμαι επιστήμονας και εκπροσωπώ την ακαδημαϊκή κοινότητα που έχει μέλη και στη Ρουμανία βέβαια και στο εξωτερικό και που είναι από αρχαιολόγοι, μαθηματικοί, φιλόσοφοι, αλλά και επιστήμονες εφαρμοσμένων επιστημών. Υπάρχει μια συνένεση στους επιστήμονες σε σχέση με τη θέση της Κομισιόν. Υποστηρίζουμε την Κομισιόν στην προσπάθειά της να αναγκάσει τη Ρουμανία να εφαρμόσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις ε, νομοθεσίες ε, έχει μεγάλη καθυστέρηση σε ορισμένα θέματα. Αλλά διαφωνούμε με τη θέση ότι η Κομισιόν θα πρέπει μόνο να περιορίσει τη δράση της σε αυτόν τον τομέα. Ε, θεωρούμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να δράσει και σε διάφορους άλλους τομείς όπου νομίζω ότι είναι της αρμοδιότητάς της για να ε, προστατεύσει την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, την ασφάλεια των πολιτών διαφόρων κρατών μελών, όχι ενός μόνο, το περιβάλλον και να δράσει υπέρ των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαίων. Καταρχάς να πω ότι ξεκινήσαμε, ξεκίνησαν αυτές οι εργασίες, αυτά τα έργα στο Ρώσια Μοντάνα, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή ενός μοναδικού, μιας μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ε, πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι θα είναι φοβερή απώλεια και πολλοί ε, διεθνείς επαγγελματικοί φορείς ζητούν να διατηρηθεί αυτός ο χώρος. Ζητάμε από την Κομισιόν να αξιολογήσει την απώλεια αυτή πολιτιστικής κληρονομιάς και να μας παρουσιάσει τους λόγους για τους οποίους θέλει να δράσει ή να μην δράσει. Τους λόγους για τους οποίους αποφασίζει κάτι. Είναι σαφές ότι το έργο αυτό είναι ιδιάζων. Είναι τελείως διαφορετικό από άλλα ε, προγράμματα, άλλα έργα, έργα Λόγω της θέσης, λόγω της, του μεγέθους και λόγω του τρόπου εκτέλεσης. Καταρχάς, η κλίμακα είναι πολύ μεγαλύτερη από άλλες ε, που προκάλεσαν και φοβερά ατυχήματα. Έχουμε 3.000 φορές περισσότερο όγκο τοξικών ε, αποβλήτων, λιμάτων μάλλον, με κιανιούχες ένωσης που είναι πολύ μεγαλύτερες από ε, ένα μεγάλο ατύχημα που έγινε στο Κολοράντο. Επίσης, θα θυμάστε το φράγμα που έσπασε στην Ουγγαρία πριν από ένα χρόνο και θα θυμάστε στις ε, τραγικές συνέπειες, ε, την απώλεια ανθρωπίνων ζώων κτλ. Το φράγμα αυτό στο Ράσο Μοντάνα θα είναι πολύ πιο ψηλό, 185 μέτρα θα είναι διπλάσιο από το άλλο φράγμα της ε, Ουγγαρίας. Επίσης η Ράσια Μοντάνα είναι πολύ πυκνοκατοικημένη και συνδέεται με το Δούναβι, είναι πολύ σημαντική τοποθεσία η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία ενδιαφέρονται και θα επηρεαστούν ενδεχομένω από το έργο αυτό και μια υποψήφια χώρα η Σερβία. Θέλουμε λοιπόν η Κομισιό να ζητήσει μια ανεξάρτητη και τίμια αξιολόγηση των κινδύνων αυτού, του έργου, που δεν υπάρχει πουθενά. Επίσης ζητάμε από την Κομισιό να ζητήσει ε, τη μελέτη και την δημιουργία σχεδίων ε, ενδεχόμενου. Επίσης, ο Καναδός ανάδοχος ε, έχει προβλέψει ένα κονδύλι 130 εκατομμυρίων ε, δολαρίων. Από, από αυτά τα έργα θα επωφεληθεί πολύ λίγο η ρουμανική κυβέρνηση και δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν αρκετά κονδύλια για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα ατυχήματα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσουμε από την Κομισιόν να, κάνουν, να κάνει υπολογισμό του ποιος θα υπομειστεί το βάρος το οικονομικό σε περίπτωση που υπάρξει ατύχημα ε, και αν τα χρήματα αυτά ε, θα είναι δημόσια ή ιδιωτικά. Γενικά, να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί με τα μέλη του Κοινοβουλίου και να γίνει μια συζήτηση για τα γενικά θέματα εδώ, όπου το κοινό, με το κοινό, την κοινωνία των πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα, μας ενθαρρύνει σε αυτό, αυτό το κύριο άρθρο, το οποίο ε, δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, όπου προβλέπεται η ε, ίδια λήψη μέτρων. Ε, είμαι είμαστε στο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αμέριστη υποστήριξή τους αν χρειαστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο επόμενο αναφέρον και σα δίνω πέντε λεφτά. Ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Ρετζούρκα και εγώ ζω στο Ρώσα Μοντάνα και είμαι αντιπρόεδρος ε, του Ιδρύματος Ρώσα Μοντάνα, του πολιτιστικού Ιδρύματος αυτού. Ζω εκεί 46 χρόνια τώρα. Και τα τελευταία 15 χρόνια η πόλη αυτή υπέστη πολλές πιέσεις εξαιτίας του γεγονότος ότι μια καναδική εταιρεία αποφάσισε ότι ήθελε ε, να προχωρήσει σε εξόριξη χρυσού στην περιοχή. Πράγμα το οποίο όμως θα οδηγήσει στην καταστροφή της Ρώσα Μοντάνα και άλλων τριών χωριών στην περιοχή. Η καναδική αυτή εταιρεία λοιπόν ξεκίνησε με την απομάκρυνση κατοίκων και αγνοεί πλήρω το γεγονός ότι εκεί υπάρχει ένας μοναδικός θησαυρό 7 χιλιόμετρα ε, ρουμανικών ε, ορυχείων υπάρχουν ε, ένα σπίτια, τα οποία έχουν φυσικά μεγάλη αξία και ακούγεται λίγο παράδοξο το γεγονός ότι το Δημαρχείο της Ρώσα Μοντάνα τελικά βρίσκεται σε ένα κτίριο το οποίο νίκει στην καναδική αυτή εταιρεία είναι ίσως ο μόνος δήμαρχος στον κόσμο που δεν δέχεται να μπει στον κατάλογο της UNESCO για πολιτιστική κληρονομιά ο Δήμος του. Όπως και άλλοι κάτοικοι της Ρώσα Μοτάν, έτσι και εγώ είμαι αγανακτισμένος με το γεγονός ότι οι τομικές αρχές μας γυρίζουν την πλάτη. Επειδή κάποιοι μπορούν ή νομίζουν ότι μπορούν να έρθουν στην περιοχή μας, να μας αγοράσουν, να αγοράσουν τα σπίτια μας, τη γη μας και μας θεωρούν εχθρούς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει διχαστεί η τοπική κοινότητα. Το σχέδιο αυτό απειλεί την περιοχή μας. Έχω τρεις ιδιοκτησίες στη βιομηχανική αυτή περιοχή που δεν θα δεχτώ ποτέ να πουλήσω στην εξορρυκτική αυτή εταιρεία. Γιατί για μένα είναι ιερό μέρος η Ρώσα Μοντάνα. Εγώ δεν θέλω να φύγω από εκεί, δεν θέλω να πουλήσω. Όπως σας είπα πρόκειται για τα σπίτια μου. Η εταιρεία αυτή καναδική θέλει να προχωρήσει στην ε, εξόριξη, πρώτα απ' όλα φτιάχνοντας ένα τεράστιο φράγμα. Και ως Ευρωπαίος πολίτης έχω μια ερώτηση. Θα μπορώ να τύχω προστασίας και να συνεχίσω τη ζωή μου στην περιοχή αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται ότι οι διοκτησίες μας ε, μπορούν να απαλωτρεθούν, να τις πάρουν αυτές οι εταιρείε και να δημιουργηθεί ένα τοξικό κλίμα στην περιοχή αυτή. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι είναι δίκαιο εμείς να χάσουμε τις ζωές μας, τις εκκλησίες μας, τα νεκροταφεία μας κλπ. κλπ οι ρουμανικές αρχές και το ρουμανικό κοινοβούλιο προσπαθούν να αλλάξουν την νομοθεσία που ισχύει όσον αφορά την εξόριξη, ώστε η απαλαιτρίωση να μπορεί να γίνει πιο εύκολα. Αν γίνει αυτό, εμείς θα πάμε στο δικαστήριο και στη Ρουμανία αλλά και στο εξωτερικό. Την εποχή αυτή είναι πολύ δύσκολο να ζει κανείς στη Ρώσα Μοντάνα. Υπάρχει τεράστια πίεση σε μας. Τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης ακόμα και αυτά ε, του έχουν κλείσει το στόμα. Δεν ε, τολμάει κανεί βασικά να μιλήσει για αυτά που συμβαίνουν στη Ρώσα Μοντάνα. Υπάρχει μεγάλη πίεση και από τα μέσα ενημέρωσης προς εμάς. Οι τοπικές αρχές συνεργάζονται στενά με την καναδική αυτή η εταιρεία εξόριξης. Και ε, μας πονάει να βλέπουμε άδεια τα σχολεία, να βλέπουμε μια πόλη που μοιάζει να έχει πληγεί από σεισμό, γιατί βλέπετε πριν από 15 χρόνια ξεκίνησε αυτή η συστηματική πολιτική της καναδικής εταιρείας να φροντίσει να γίνουμε όλοι πιο φτωχοί, πιο φτωχοί να αναγκαστούμε να φύγουμε, να μην μπορούμε να προχωρήσουμε σε καμία επιχειρηματική δραστηριότητα, να μην μπορεί κανείς να φτιάξει κάτι καινούριο. Κάθε φορά που προσπαθούσε κάποιο να το κάνει αυτό, η καναδική εταιρεία έδινε περισσότερα χρήματα και τον ανάγκασε να φύγει. Στόχος της είναι να αποκτήσει όλα τα σπίτια, όλη τη γη, να αγοράσουν τα πάντα, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν με το σχέδιό τους. Αν δεν απατώμε μάλιστα το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει λάβει αίτηση ώστε να γίνει πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO η Ρώσα Μοντάνα. Βέβαια φοβάμαι ότι μας μένει πολλής δρόμος μέχρι να το πετύχουμε αυτό. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε μια στιγμή. Θέλω να σας δώσω τον τουριστικό οδηγό που έχουμε ετοιμάσει στη Ρώσα Μοντάνα. Είναι ένα δώρο από μας σε εσά. Σε το δεύτερο αναφέροντα. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει το λόγο, εκπροσωπείται εδώ. Δεν με να πω το όνομά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ του αναφέροντες γιατί παρουσιάσαμε με πολύ καλό τρόπο το πρόβλημα. Έχει υποβληθεί αυτή η αναφορά ήδη όταν, όταν ήμασταν σε αρχική φάση του έργου. Προτού δηλαδή τα βασικά έγγραφα ε, συνταχθούν όπως η μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου κτλ. Χωρίς αυτά τα έγγραφα είναι αδύνατον εμείς να αποφασίζουμε ότι υπάρχει παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το γεγονός ότι είμαστε πολύ νωρίς στη διαδικασία μας επιτρέπει όμως από πλευράς Κομισιόν να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες από τις ρουμανικές αρμόδιες αρχές για το κατά πόσον η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία γίνεται σεβαστή και ιδίως η οδηγία για τον τρόπο εξόριξης. Οι ρουμανικές αρχές προς τις οποίες απευθυνθήκαμε μας έχουν δώσει περαιτέρω πληροφορίες τις οποίες επεξεργάζεται και θα διαβιβάσει οι υπηρεσίες ε, της Κομισιόν. Η Κομισιόν έχει απαντήσει στους θα απαντήσει μάλλον ε, στους αναφέροντες μετά από την επεξεργασία όλων αυτών των στοιχείων. Θα ήθελα να αναφερθώ καταρχάς στον πρώτο, να απαντήσω μάλλον στον πρώτο αναφερόμενο. Παραμένω στην αρχική θέση της Κομισιόν, δηλαδή ότι παρότι καταλαβαίνουμε την κοινωνικονομική, ιστορική και πολιτιστική σημασία του προβλήματος, η τελική απόφαση δεν είναι δική μας, αλλά των αρμόδιων ρουμανικών αρχών. Εμείς θα ζητήσουμε ανάλυση των στοιχείων. Αλλά δεν είναι εξουσία δική μας, δεν είναι αρμοδιότητα δική μας να αποφασίσουμε, αλλά του κράτους μέλους. Ε, Ξεκινάει η συζήτηση. Ο κύριος Μποσινάρου. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαίρομαι για την προσπάθεια και για το ζήλο με τον οποίο οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις από τη Ρουμανία καταπολεμούν αυτό το έργο, το εξορρυκτικό οι οικονομικοί φορείς της ε, Ρουμανίας, οι απλοί ερευνητές, ε, διάφοροι παράγοντες ενεπλάκησαν και διαμόρφωσαν αυτή τη θέση και πολεμούν αυτόν τον πόλεμο. Ανάμεσα, ένας πόλεμος μεταξύ της φύσης και της βιομηχανίας. Ξέρετε ότι ο πρόεδρος της Ρουμανίας είναι ένθερμος θειασότης αυτού του έργου παρά τα όσα λέει το Σύνταγμα. Θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτά που είπε η Κομισιόν. Η Κομισιόν λέει ότι με βάση τις πληροφορίε που έχει, αυτή η εταιρεία της Ράσα Μοντάνα ε, θα δώσει 150 ε, εκατομμύρια ευρώ για έργα συντήρησης, εποπτείας των ε, δεξαμενών λιμάτων που θα χτιστούν. Έχουμε ένα τεράστιο, ένα γιγαντιαίο έργο. Είναι, θα είναι το μεγαλύτερο χρυσορυχείο στον πλανήτη αυτό. Είναι ένα έργο το οποίο απαιτεί την εξκαφή πάνω από 5.000 εκατομμύρια 5 δισεκατομμύρια δηλαδή τόνους πολύ περισσότερο από ό,τι χρησιμοποιεί μέχρι στιγμής ε, η υπόλοιπη βιομηχανία. θα χρησιμοποιούνται 13.000 τόνοι κυανιούχων ενώσεων το χρόνο. Δηλαδή 13.000 περισσότερο το χρόνο. Μέσα σε μία περίμετρο 1.200 εκταρίων θα δημιουργήσει ένα τεράστιο κρατήρα που θα είναι ορατός από τη σελήνη. Θα έχει διάμετρο 8 χιλιόμετρα και η μεταφορά των αποβλήτων που θα προκύψουν από τη χρήση των εκρηκτικών, γιατί θα χρησιμοποιήσουν 10 τόνους δυναμίτη κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο. Αυτά τα απόβλητα θα μεταφέρονται με φορτηγά 150 τόνων που θα γιγαντώσουν την ε, μόλυνση, τη ρήπανση, καθώς και τις, ε, τους κραδασμούς που θα δημιουργήσουν προβλήματα στο φράγμα. Τώρα αυτά είναι όλα τεχνικά στοιχεία, γιατί θέλω να ε, κρούσω τον κόδωνα στην, στην Κομισιόν για το καταστροφικό, την καταστροφική επίπτωση που θα έχει στο περιβάλλον. Αυτές οι δεξαμενές αποβλήτων θα είναι τεράστιες και θα έχουν μέσα κιανιούχες ενώσεις. Το βασικό στοιχείο θα είναι κιάνιο, δηλαδή και βαριά μέταλλα για να καταλάβετε το μέγεθος αυτού προβλήματος και τους τεράστιους κινδύνους που αφορούν όχι μόνο την ασφάλεια της Ρουμανίας αλλά την ασφάλεια και των γειτονικών χωρών. Να σας υπενθυμίσω αγαπητοί συνάδελφοι ότι το 1993 ένα πολύ πολύ μικρότερο ατύχημα έγινε στις ΗΠΑ στο Κολοράντο. Το 1995 έγινε αντίστοιχο ατύχημα στη Γουιάννα. Το 1998 στο Κυργιστάν και το 2000 στο Μπαμάρε στην Ρουμανία. Το ατύχημα αυτό θεωρήθηκε από τα ουγγρικά μέσα ενημέρωση ως δεύτερο Τσερνομπίλ και προέκυψε από την διαρροή α, χιλίων τόνων κιανίου και κιανιούχων ενώσεων που κατέστρεψαν την χλωρίδα και την πανίδα του Τίσαν, του ποταμού Τίσαν. στην ε, περίπτωση του Ράσο Μοντάν θα έχουμε πολύ περισσότερο, πολλαπλάσιο ε, κιάνιο. Και το φράγμα που θα προκύψει θα είναι 185 μέτρα. Θα πρέπει να κρατήσει για πάντα, μέχρι το τέλος, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Η καναδική εταιρεία, στη, μέσα στη μεγάλη αυτή α, γενεοδορία της, θα δώσει μάλλον 150 εκατομμύρια για τη συντήρηση αυτού του φράγματος. Σκεφτείτε τι έγινε πέρυσι στην Ουγγαρία με το ατύχημα, το οποίο προκλήθηκε από την έκκληση λασπόνερων, ε, μολυσμένων, 700.000 τόνων. Επιβλήθηκε πρόστιμο, αλλά ήταν αστείο το πρόστιμο. Ενώ τώρα στην περίπτωση της Ρέσο Μοντάνα έχουμε μια οικολογική βόμβα. Θα την διαχειριστούμε μόνο με 150 εκατομμύρια ευρώ εμείς ε, τότε επιβάλαμε στην Ουγγαρία 500 εκατομμύρια ευρώ στους, α, στους Ούγγρους ως πρόστιμο για την ζημιά που υποστήκαμε. Και εδώ δηλαδή για ένα πολύ μεγαλύτερο έργο διατίθενται μόνο 150 εκατομμύρια. Τι θα γίνει όταν γίνει καταστροφή. Η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν νομίζω ότι μπορεί να αποφέρει τις ευθύνε της. Και θα ήθελα να σας πω εν κατακλείδη το εξή. Συμφωνώ ότι αυτά τα νούμερα τα οποία κυκλοφορούν ε, μοιάζουν ενδιαφέροντα. Αλλά θεωρείται ότι το κόστος ε, εκμετάλλευσης και, ε, με βάση μία αυστραλέζικη εταιρεία θα είναι 600 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ κάποιοι Αμερικάνοι λένε ότι θα είναι 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Κοιτάξτε τη διαφορέ των νούμερων εδώ. Εγώ υποστηρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δράσει και να παρέμβει. Και τα λεφτά που προέρχονται από το χρυσό εξαγοράζουν τα σπίτια των φτωχών, ε, αγοράζουν πολιτικούς, ε, βάζουν τις κατάλληλες διαφημίσεις, αγοράζουν ακόμα και κυβερνήσεις. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έχουν μια στεναρή στάση με βάση την νομοθεσία. Και κάτι άλλο, Κομισιόν. Εδώ δεν ασχολούμαστε μόνο με την οδηγία που αφορά την εξορρυκτική βιομηχανία. Εδώ μιλάμε για τα υπόγεια νερά και τη σχετική οδηγία, για την οδηγία για την ποιότητα του αέρα. Θα πρέπει να έχετε μια ε, στρατηγική θεώρηση και επίσης μια μελέτη για τις επιπτώσεις αυτής τη οικολογική βόμβας. Σας καλώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβετε δράση. Δεν πρέπει να δράσετε εκ των υστέρων ή αφού γίνει η δολοφονία αυτή του περιβάλλοντος. Μην με αναγκάζετε να δειχτώ, να γίνω πάρα πολύ αυστηρή. Αλλά αν ο καθένας από εσά μιλάει 10 λεπτά, δεν θα μιλήσουν όλοι. Σας παρακαλώ, εγώ θέλω να δώσουμε χώρο και χρόνο στους αναφέροντες να μιλήσουν περισσότερο. Η κυρία Ταμπάτζη, ή ο κύριος Ταμπάτζη μάλλον. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Πιστεύω ότι όσοι πήραν το λόγο πριν από μένα έχουν ε, ήδη εξηγήσει ότι υπήρξαν ε, και άλλα ατυχήματα που έγιναν ε, κατά το παρελθόν, εκείνο της Βαγιαμάρα για παράδειγμα, όπου έχασαν τη δουλειά τους 10.000 άνθρωποι και που θα πάρει χρόνια βέβαια να ξαναφτιαχτεί η περιοχή. Μέχρι σήμερα κανένας ε, Ούγγρος πολίτης δεν έχει πάρει την παραμικρή αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστησαν. Ως μέλος και της Επιτροπής Περιβάλλοντος θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε μερικά σημαντικά νομίζω πράγματα. Πρώτα απ' όλα, εγώ χαίρομαι που υπάρχει η ανακοίνωση της Επιτροπής, αλλά νομίζω ότι είναι ανεπαρκής. Θέλω λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποια γεγονότα. Χρησιμοποιείται η τεχνολογία στην Ευρώπη, στη Σουηδία, στη Φιλανδία. Χρησιμοποιούν όμως μια εντελώς διαφορετική τεχνολογία Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να ρωτήσουμε όσον αφορά την εξόριξη. Γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την τεχνολογία απομόνωσης των κοινούχων ενώσεων και εκεί όπως χρησιμοποιείται αυτή στην Σουηδία και στη Φιλανδία. Ε, τέτοιες τεχνολογίες προστατεύουν το περιβάλλον. Ενώ εδώ με το σχέδιο αυτό έτσι όπως προβλέπετε δεν υπάρχουν τέτοιες εγγύσεις. Κάτι άλλο στο οποίο θέλω να πιστήσω την προσοχή σας είναι η οδηγία REACH. Εδώ βέβαια δεν πρόκειται να σας τη διαβάσω. Θα κυκλοφορήσω όμως, θα σας μοιράσω την παράγραφο η οποία όμως λίγο πολύ λέει εξή Εάν μέσα στην ίδια τεχνολογία και μέσα στο ίδιο σχέδιο ξέρουμε ότι υπάρχει ένα άλλο το οποίο ε, ρηπαίνει λιγότερο το περιβάλλον, τότε η τεχνολογία αυτή, η κλειστή για τις καινούχιες ενώσεις, στην οποία αναφέρθηκα πριν που χρησιμοποιείται στη Σουηδία και την Φιλανδία, πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί άλλες εταιρείε η Αυστραλία χρησιμοποιεί αυτή τη τεχνολογία και δεν ε, την χρησιμοποιούμε σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν βέβαια διαφορές ανάμεσα στη Σουηδία, τη Φιλανδία και την Ρουμανία. Και αυτή είναι ότι στη Σουηδία και στη Φιλανδία οι παραβιάσει της οδηγία REACH τιμωρούνται πάρα πολύ αυστηρά, ενώ στην Ρουμανία παραβιάσεις τέτοιες δεν τιμωρούνται με την ίδια αυστηρότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή της Ρουμανίας στο γεγονός ότι στην Ρουμανία δεν υπάρχουν ε, ποινικέ κυρώσει, μόνο διοικητικέ. Εάν δηλαδή η επιχείρηση αυτή παραβιάσει τις ε, διατάξεις της οδηγίας REACH θα πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες κυρώσεις έτσι ώστε οι υπεύθυνοι να διώκονται βάσει του ποινικού δικαίου. Η ευθύνη για το περιβάλλον είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να απευθυνθεί στις ρουμανικές αρχές προκειμένου να αναγκάσουν την καναδική εταιρεία να έχει εγγύηση αρκετά μεγάλη, να δώσει αρκετά μεγάλη εγγύηση που να μπορεί να καλύψει οτιδήποτε κινδύνους προκληθούν και οποιοδήποτε ατύχημα προκύψει από την ε, λειτουργία αυτή. Επί έξι πρέπει να υπολογίζουμε ε, τα χρήματα τα οποία προτείνονται σήμερα. Το σχέδιο αυτό της Ρώσα Μοντάνα περιβαλλοντικά ελοχεύει τέτοιους κινδύνους που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αρκεστεί έτσι ηθικά ε, στα όσα προσφέρονται και να στηρίξει αυτό το σχέδιο. Γιατί υπονομεύει το περιβάλλον. Δεν πρέπει να συνεχιστεί. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε. Θέλω εδώ να χαιρετήσω όλους τους ε, ε, όσους πήραν το λόγο από τους αναφέροντες και όλα τα μέλη της Επιτροπής που πήραν το λόγο. Δεν θέλω να επαναλάβω τέτοια και τα ίδια, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι φυσικά και πρέπει να εγγυθούμε την προστασία των πολιτών και στο μέλλον. Είναι προστασία ολόκληρη της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε νέα τέτοια καταστροφή. Τη στιγμή που γνωρίζουμε τις συνέπειες μπορεί να έχει μια καταστροφή πολύ μικρότερη που είχαμε πρόσφατα. Στην περίπτωση αυτή του ρωμανικού σχεδίου θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη καταστροφή. Στην Ουγγαρία ξέρετε τι έγινε και πώς καταστρέφτηκε η πανίδα και η χλωρίδα του ποταμού Τίσα και που 10 χρόνια χρειάζονται για την αποκατάσταση της περιοχής. Το επίπεδο της ε, ρήπανσης ξεπέρασε κατά 110 τα αποδεκτά όρια. Εδώ μιλάμε για πολύ μεγαλύτερες καταστροφές και ξέρουμε ότι η άδεια για να δοθεί στην ε, καναδική αυτή εταιρεία έχει πάρει 10 χρόνια. Υπάρχουν ένα σωρό μη κυβερνητικέ οργανώσει που παρεμβαίνουν, γιατί ακριβώ υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι. Έτσι λοιπόν, πολύ απλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το τι έχει συμβεί στο παρελθόν και να κάνουμε σαν να μην ξέρουμε τίποτα. Το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει μέτρα ώστε να απαγορευτεί η χρήση της τεχνολογίας αυτής για τις κιανούχες ενώσεις. Τελικά τι έκανε η Επιτροπή, τίποτα. Πρέπει να απαγορευτεί η τεχνολογία αυτή που είναι επικίνδυνη και να χρησιμοποιηθούν άλλε τεχνολογίε τι οποίε επιτρέπει, επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που δεν είναι τόσο επικίνδυνε. Χρειάζεται λοιπόν μια πρωτοβουλία. Νομίζω ότι είναι μεγάλη παράληψη να μην έχει κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την απόφαση που πήρε πέρυσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρουμε επίση ότι υπάρχουν πολλέ διαμαρτυρίε από του πολίτε στη Ρουμανία. Υπάρχει μια διαδικασία με συλλογή υπογραφών μέσω του διαδικτύου που έχει πάνω από 17.000 υπογραφές. Ε, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι πρέπει με τι άλλο να δώσουμε σημασία στις προσφυγές που κάνουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αλλιώς θα εξαφανιστούν αξίες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι και οι αναφέροντες. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, ούτε να βάζουμε το κεφάλι στη γη και να κάνουμε πως δεν βλέπουμε την καταστροφή αυτή που προαναγγέλλεται η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι αποδεκτή. Η Επιτροπή λέει ότι είμαστε στην αρχή της διαδικασίας ε, παραχώρησης της άδεια και θα δούμε τι θα γίνει στη διαδικασία. Ε, όχι, γιατί εγώ φοβάμαι ότι θα υπάρξει μια καταστροφή την οποία, σχετικά με την οποία δεν θα μπορούμε να κάνουμε επίση Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να υποβάλει πρόταση με την οποία να απαγορεύεται η τεχνολογία αυτή και ανούχων ενώσεων και να απαγορευτούν αυτές όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας τους Ρουμάνους αναφέροντες. Τους ευχαριστώ για την παρουσίαση που έκαναν. Να προσθέσω και εγώ δύο λόγια για την ε, κατάσταση στη Ρώσια Μοντάνα και πρώτα να σας θυμίσω κάποια βασικά στοιχεία Δηλαδή, η αναφορά αυτή αφορά ένα έργο. Έργο είναι μόνο, δηλαδή επί χάρτου. Δεν έχει αρχίσει τίποτε. Μόνο στα σχέδια βρίσκεται. Δεν γίνεται δηλαδή ε, εξόριξη εκεί, δεν υπάρχει μεταλλείο χρυσού εκεί είναι μόνο στα χαρτιά το σχέδιο. Η πρόθεση έναρξης εξορυκτικής δραστηριότητας εκεί είναι παλιά, από το 1994. Και το Δεκέμβριο του 2004 η εταιρεία αυτή έδωσε κάποιους πόρους, έκανε την αίτηση και τα προηγούμενα 7 χρόνια δηλαδή, από το 2004, αυτή η πρόθεση έργου συζητείται. Δεν έχει αρχίσει λοιπόν τίποτε εκεί. είναι στις συζητήσεις. Και όλα τα άλλα στοιχεία που αφορούν το θέμα αυτό, οι αντιδράσεις των ρουμανικών αρχών στην έκφραση αυτή των, ε, του ενδιαφέροντος, όλα αυτά είναι ε, διαθέσιμα ε, στο διαδίκτυο και όλοι έχουν πρόσβαση τα έχω αυτά να τα δώσω και στον συνάδελφο Μποστινάρο, ο οποίος εκτός μικροφώνου έκανε μια παρατήρηση. Να σας τη δώσω την έκθεση κύριε Μποστινάρο, άμα θέλετε να τη διαβάσετε, τι άλλο πια να κάνω. έχουν γίνει πολλές δημόσιες συζητήσεις στη Ρουμανία. Να μην κάνουμε διάλογο. Ε, λοιπόν, ε, συνεχίζει ο κύριο Πρέντα Αυτές λοιπόν οι αμέτρητες συζητήσεις, ε, ε, κάποιες από αυτές τουλάχιστον, συνδιοργανώθηκαν ή οργανώθηκαν από τις ρουμανικές αρχές. Αυτοί που θέλουν το έργο απάντησαν στις ανησυχίες ε, της κοινή γνώμης, έδωσαν κάποιες εκτιμήσεις και οι επιπτώσεις περιβαλλοντικής περιβαλλοντικές επιπτώσεις ε, παρουσιάστηκαν. Η αναφέροντες τώρα αναφέρονται σε πολλές ε, νοσιακές οδηγίες που υποτίθεται ότι παραβιάστηκαν από το έργο της στη Ρώσια Μοντάνια. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα, γιατί πώς είναι δυνατόν να παραβιάζονται οι οδηγίες αυτές αφού το έργο δεν άρχισε καν. Ένα σχέδιο επιχάρτου δεν μπορεί να παραβιάσει καμία οδηγία. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι χρονοδιάγραμμα ακολουθεί το πρόγραμμα. Τώρα είναι στη διερευνητική και όχι στην επιχειρησιακή φάση του το πρόγραμμα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν τα συζητάμε αυτά. Από την άλλη, είναι κρίμα που έκαναν όλο το δρόμο να έρθουν μέχρι τις Βρυξέλλες οι αναφέροντες για να διαπιστώσουν ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε το Κοινοβούλιο δεν έχουν την ε, δυνατότητα να σταματήσουν ένα έργο φαντάζομαι ότι αυτό θα μπορούσατε να το είχατε πληροφορηθεί πιο εύκολα. Δεν το ξέρατε. Πάντως, οι ρουμανικές αρχές έχουν την ε, αρμοδιότητα να αποφασίσουν τέτοια πράγματα. Και τα προηγούμενα χρόνια δεν ελήφθη καμία απόφαση, τα προηγούμενα 7 χρόνια. Έχουν γραφτεί δεκάδες χιλιάδες ε, έγγραφα, τα οποία υποβλήθηκαν ως μέρος του έργου αυτού, αλλά απόφαση ακόμα δεν ελήφθη. Από την άποψη της ευρωπαϊκής κοινή γνώμης, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι τώρα η εταιρεία που υπέβαλε το έργο, όπως και οι ρουμανικές αρχές, εξετάζουν πώς θα σεβαστούν την ενωσιακή νομοθεσία. Τώρα υπάρχει ένας συνασπισμός ε, αυτών που αντιδρούν στο έργο και κάνουν πολύ επιθετικό λόμπι και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ε, Ρουμανική Κοινή Γνώμη και έχουν εφεύρει την αντίληψη ότι οποιαδήποτε μορφή χρήσης τεχνολογίας στην εξόριξη των κοινούχων ενώσεων απαγορεύεται. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι τεχνικές λύσεις ε, που πρέπει να δώσει η ε, μεταλλευτική εταιρεία θα ακολουθήσουν την αυστηρή νομοθεσία της Ένωσης. Κανείς δεν λέει ότι αρνείται να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αντιθέτως, έχουν πει δημοσία ότι θέλουν να ακολουθούν όλα τα πρότυπα ασφαλείας. Και αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στο διαδίκτυο και όποιος θέλει μπορεί να τα κατεβάσει. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζήτησε ε, ειδικέ εγκαταστάσεις για να αντιμετωπίζει να, ούτε, να μην, ε, η, η συγκέντρωση των κυανιούχων ενώσεων να μην υπερβαίνει τα 3 ppm στις λίμνες αυτές ε, από βλήτων από την εξορυκτική βιομηχανία. Και αυτά υπάρχουν. Ενώ οι ε, ενάντια στο έργο λένε ότι κανείς δεν νοιάζεται για αυτά. Οι δημόσιες συζητήσεις δείχνουν το αντίθετο όλες οι ανησυχίες των αναφερόντων και από του κυρίου Μποστινάρου και των άλλων συναδέλφων, όλες αυτές οι ανησυχίες έχουν μελετηθεί, έχουν ληφθεί υπόψη. Τώρα, εις ό,τι αφορά τις ε, οικονομικές ε, εγγύησεις, και αυτό το θέμα αξιολογείται, εκτιμάται ε, και βεβαίως το σημαντικό είναι αυτή η ανησυχία που εξέφρασε και ο κύριος Μποστινάρου. Τέλος, να πω ότι λυπάμαι, διότι η όλη συζήτηση για το Ρώσια Μοντάνια έχει εκτροχιαστεί προς θέματα που δεν έχουν να κάνουν με τη Ρώσια Μοντάνα και τις αναφορές των διακεκριμένων εδώ αναφερόντων. Ο κύριος Ποστινάρου, για παράδειγμα, ε, μίλησε για το Ρουμάνο πρόεδρο και τη στάση του. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Ο κύριος Ποστινάρου μίλησε για κάποιους Ρουμάνους πολιτικούς που έχουν εξαγοραστεί, εξονημένους. Τι είναι αυτά, δεν έχουν σχέση. Αν σκεφτούμε την προηγούμενη 7 ετία και τι συνέβη, θα έλεγα ότι αυτοί που είναι κατά του έργου μπορεί να έχουν εξαγοραστεί από κάποιον. Μην μπαίνουμε σε πολιτικές ε, τέτοιες ε, συζητήσεις. Όχι, καλό θα ήταν να είχατε παρέμβει και όταν μίλησε ο κύριος Μποστινάρου, λέει ο κύριος Πρέντα. Ε, την ίδια στάση έπρεπε να τηρήσετε και όταν μίλησε ο κύριος Μποστινάρου. Εγώ δεν ε, υπερασπίζομαι τον κύριο Μποστινάρου, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Πρέντα, να τελειώσω λέγοντας ότι έχω και μία ερώτηση για την επίσκεψη στη Ρουμανία. Ξέρω, κάποιος πρότεινε να συζητήσω με τις αναφορές αυτές όταν θα πάμε στη Ρουμανία. Αναρωτιέμαι λοιπόν, γιατί συζητάμε σήμερα λοιπόν και γιατί θα πρέπει και τον άλλο μήνα να το ξανασυζητήσουμε. Δηλαδή τι θα γίνει, κάθε μήνα θα το συζητάμε, είμαστε υποχρεωμένοι. Τι είναι αυτό, τι διαδικασία είναι αυτή. Αφού γίνεται συζήτηση σήμερα, γιατί πρέπει όταν θα πάμε στο Βουκαγουρέστι να ξανασυζητήσουμε τα ίδια πράγματα, οι ίδιοι άνθρωποι. Α μα πει ίσω ο κύριο Μποστινάρου που είναι συντονιστή τη Σοσιαλιστική Ομάδα ή να μου εξηγήσετε εσεί κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να σα εξηγήσω. Θα δούμε όταν θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα για την επίσκεψη στη Ρουμανία τι προτάσεις για ποιες θέσεις θα πρέπει να επισκεφτούμε ως Επιτροπή Αναφορών. Θα έχετε όμως πολύ σύντομα το τελικό πρόγραμμα. Προηγείται η κυρία Βαλεάν παρακαλώ. Αλλά θα, κάνω έκκληση αν μπορείτε σύντομα γιατί έχουμε δύο ακόμη ε, καταγγέλλοντες που θα παρουσιάσουν τα δικά του ζητήματα και στις 11 περιμένουμε την Πολωνή διαμεσολαβήτρια. Ευχαριστώ. Oh, thank you, Um, Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά για αλλαγή. Έχουμε την καναδική εταιρεία, έχουμε τη Ρουμανία στην οποία φτιάχνεται το σχέδιο αυτό. Όμως το θέμα του περιβάλλοντος δεν έχει σύνορα και γι' αυτό εμείς συζητάμε εδώ το θέμα των απειλών στο περιβάλλον. Είμαι μέλος βέβαια και της Επιτροπής Βιομηχανίας. Οπότε πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι κάτι εύκολο. Μία χώρα μέλος πρέπει να κάνει την επιλογή κατά πόσο δέχεται ή όχι βιομηχανικά σχέδια. Υπάρχουν τόσο πολλές ε, βιομηχανίες τις οποίες μπορεί να προκύψει ένα ατύχημα ή να υπάρξει πρόβλημα για το περιβάλλον. Το ερώτημα δηλαδή, το δίλημα που έχουμε είναι να έχουμε βιομηχανία ή να μην έχουμε. Αυτό το δίλημα τίθεται στις χώρες μέλη. Αλλά γι' αυτό έχουμε και οδηγίες. Ευρωπαϊκές οδηγίες που καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια προκειμένου να λειτουργήσει μια βιομηχανία. Άρα είναι φιλοσοφικό το ζήτημα. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε ένα τέτοιο σχέδιο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά πόσο υπάρχει παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου ή όχι. Κατά τη γνώμη μου όχι, αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που πρέπει να απαντήσει, έτσι θα είναι ευτυχείς όλες οι πλευρές. very Θα είμαι πολύ σύντομη. Θέλω να υπογραμμίσω ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική αναφορά. Και θα έλεγα στον κύριο Μπρέντα, γιατί νομίζω ότι προσβάλλατε τους αναφέροντες κύριε Μπρέντα αυτά που λένε είναι σωστά και αυτό που λέτε εσείς, το είπατε και εσείς ότι δεν είναι παράνομο να πούν αυτά που είπανε. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες είναι πάρα πολύ αυστηροί και γι' αυτό οι αναφέροντες εκφράζουν το φόβο τους ότι δεν θα τηρηθούν οι ευρωπαϊκοί κανόνες και πρέπει να είμαστε ευγνώμονε προς τους αναφέροντες που έρχονται και μας παρουσιάζουν την αναφορά τους. Εγώ είμαι που έχουμε αυτά τα στοιχεία και μπορούμε και τα συζητάμε. Και πρέπει να σας πω ότι αισθάνθηκα κάπως άσχημα για αυτά που είπατε για τη δουλειά τους. Ήθελα να το έχω πει. Είναι όντως ένα από τα δύο πιο σημαντικά θέματα που έχουμε όσον αφορά τη Ρουμανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, επομένως, ε, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και στους ε, αναφέροντες και μία προς την Επιτροπή. Αν οι αναφέροντες θέλουν να ακυρώσουν αυτή την εξόριξη χρυσού στη συγκεκριμένη περιοχή ή όχι, δεν έγινε σαφές και στην Επιτροπή αν θεωρεί ότι το θέμα αφορά μόνο τη Ρουμανία ή μήπω αφορά και τις γειτονικές χώρες. Κάτι που αναφέρεται σε μία από τις δύο αναφορές, Σε ό,τι τουλάχιστον αφορά τη χρήση του, του, φράγματος. Γιατί αν είναι έτσι τότε το ζήτημα δεν είναι απλά της Ρουμανίας, το ζήτημα είναι και της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα περίμενα μια απάντησή σας. Σε ό,τι αφορά την πρόταση των καταγγελόντων να ε, γίνει μια ανεξάρτητη επιτροπή που θα εξετάσει όλα αυτά τα ζητήματα περιβαντολογικά αρχαιολογικά πολιτιστικά δηλαδή κλπ νομίζω ότι θα έπρεπε να τη σκεφτεί πολύ σοβαρά η κομισιόν. ευχαριστώ. Πολύ σύντομος θα είμαι. Θα μιλήσω γενικά, χωρίς να παραβλέπω το βάσιμο της αναφοράς. Θα ήθελα να μιλήσω κυρίως όμως για τη λειτουργία της Επιτροπής Αναφορών μας. Μήπως ε, μας έφτασε αυτό το σημείο πολύ νωρίς, γιατί να μην περιμένουμε λιγάκι να υπάρξει μια απόφαση ή να γίνει μια μελέτη αντικτύπου, αλλιώς θα μας πλημμυρίζουν μονίμως με διάφορα έργα, με διάφορα σχέδια τα οποία ε, θα προκύπτουν. Μήπως ε, καλύτερα θα ήταν να περιμένουμε περισσότερο πριν αποφανθούμε να, προχωρήσω λίγο τα έργα. Είναι πολύ νωρί να αποφανθούμε, χωρί να αμφισβητώ το βάσιμο τη αναφορά. Αλλά με, το, με βάση τον τρόπο λειτουργία τη Επιτροπή μα, νομίζω ότι ασχολούμαστε με το θέμα πολύ, πολύ νωρί. Ε, προεδρεύω, δεν μπορώ να έχω άποψη σε αυτή τη φάση. Ε, πολύ σύντομα, αν θα ήθελαν οι καταγγέλλοντε και η Επιτροπή να απαντήσουν ή να κλείσουν αυτή τη συζήτηση για την ώρα. Ε, και έχω να σας κάνω και μια ανακοίνωση μετά. Θα ήθελα να πω στον κύριο Πρέντα ότι είναι αλήθεια ότι το, τα έργα δεν έχουν αρχίσει ακόμα. Αλλά όμως είναι τμήμα των έργων που έχει προσχεδιάσει η ρουμανική κυβέρνηση. Είναι αλήθεια. Βασίζονται εκεί, σε αυτό το έργο. Τσεκάρετε το. Θα δείτε ότι έχω δίκιο. Όταν ο Πρωθυπουργό, ο κύριος Μποκ, έχει, έκανε την ε, δημόσια δήλωση και είπε ότι αυτό το έργο είναι προτεραιότητα της ε, κυβέρνησης και του κυβερνητικού προγράμματος, το άκουσα αυτό, το είπε, το άκουσα με τα αυτιά μου. Και το έργο αυτό, η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια. Μπορείτε να διαρωτηθείτε γιατί πήρε 15 χρόνια για να ξεκινήσει. Γιατί τέσσερα ή πέντε διαφορετικά υπουργικά συμβούλια δεν είχαν το θάρρος να εγκρίνουν τη δρομολόγηση αυτού του έργου. Γιατί αυτό που ενέκριναν οι τοπικές αρχές ήταν εναντίον του νόμου. Πολλοί έκαναν μήνυση εναντίον της απόφασης της ε, τοπικής αρχής. Ο κόσμος θέλει να ζήσει ελεύθερα εκεί πέρα, ήσυχα στη Ράσο Μοντάνα, όπω ζει κανεί στο Βουκουρέστι ή εδώ στι Βρυξέλλε. Θέλουμε να μα αντιμετωπίσετε σαν Ευρωπαίου πολίτε. Αλλά στη Ράσο Μοντάνα παραβιάζεται ο νόμο και αυτό γίνεται εδώ και 15 χρόνια. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και έτσι κλέβετε χρόνο ουσιαστικά τι επόμενε αναφορές. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Στη γραπτή μας απάντηση προσπαθήσαμε να ξεκαθαρίσουμε τρία πράγματα. Καταρχάς, ότι το έργο αυτό, λόγω της θέσης και του μεγέθους, ε, είναι, αποτελεί δική του κατηγορία. Είναι καμία σχέση με άλλα έργα αντίστοιχα. Καμία σχέση. Είναι ιδιάζων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, ιδιαίτερη προσοχή να δώσουμε σε αυτό το έργο. Να το, να το δούμε χωριστά, ανεξάρτητα από, από όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερον, δεν έχει αξιολογήσει κανένας με αξιόπιστο και ανεξάρτητο τρόπο τους κινδύνους. Δεν υπάρχει καμία έκθεση που να είναι πλήρης και που να την έχει συντάξει άνθρωπος του οποίου η αξιοπιστία δεν αμφισβητείται. Όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί και έχουν συντάξει εκθέσεις έχουν συμφέροντα. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων λοιπόν. Θα πρέπει η Επιτροπή Αναφορών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει μια ανεξάρτητη έκθεση από ανθρώπου δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν συμφέροντα, ίδια συμφέροντα. Το μέγεθο τώρα του έργου είναι τέτοιο που σε περίπτωση που γίνει ατύχημα θα είναι τεράστιο. Δεν έχουμε αξιολόγηση αυτών των ενδεχόμενων ατυχημάτων. Εμείς είπαμε στην Κομισιόν ότι και το λέει και η επιστολή της Κομισιόν ότι σε αυτή την περίπτωση όταν υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι υπάρχει η αρχή της πρόληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να εφαρμοστεί. Ειδικά όταν τα έργα αυτά ενέχουν τρομερούς κινδύνους. Και εμείς ζητάμε να σταματήσει προσωρινά το έργο μέχρι να γίνει προσεκτική αξιολόγηση των κινδύνων. Να υπάρξουν επίσης και να δημιουργηθούν και σχέδια για πάνε ενδεχόμενο που θα αντιμετωπίζουν κάθε κίνδυνο. any, any Ευχαριστώ. Η Κομισιόν σχόλια. Ε, λάβαμε δύο ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα γρήγορα. Πρώτη ερώτηση αφορά τη διεθνή διάσταση του έργου. Με βάση αυτά που γνωρίζω το έργο είναι αρκετά μεγάλο ώστε να υπόκειται στη Σύμβαση για την, ε, τον έλεγχο περιβαλλοντικών επιπτώσεων ε, και θα πρέπει σε αυτό να συμμετέχουν και οι γειτονικέ χώρες. Δεύτερη ερώτηση. Ε, σύσταση ανεξάρτητη ανεξάρτητης επιτροπής ε, για να δει θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, κοινωνικά κλπ. Ε, ως μέλος της ε, Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος δεν νιώθω άνετα να παρουσιάσω αυτό το θέμα. Τώρα θα το θέσω στους αρμόδιους συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα επανέλθω με την απάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν ανακεφαλαιώσουμε. Ενημερώνω ότι νωρί σήμερα το πρωί η γραμματεία έλαβε ένα email με την επίσημη θέση της Ρουμανικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας και για το σημερινό μας θέμα και για την αναφορά υπαριθμών 27 για τους ανεμόμυλους που θα μας απασχολήσουν το απόγευμα. Η επιστολή θα είναι στην διάθεσή σας αφού μεταφραστεί το συντομότερο. Τέλος, αυτό που απάντησε η Κομισιόν είναι να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά, περιμένουμε τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη διερευνητική μας επίσκεψη και περιμένουμε να δούμε τι θα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά, ε, δηλαδή τι θα πει μετά από τον έλεγχο από αυτή την ανεξάρτητη επιτροπή ή ομάδα. Εντάξει, ευχαριστούμε. Πάμε στο επόμενο, που δεν είναι το 16, αλλά το 17, γιατί ήρθε η αναφέρουσα. Η κυρία Σίλα Έλλης θα μιλήσει, εξ ονόματος οργάνωση κάτι και κατά τοξικού χώρου ταφής, αποβλήτων. Ορίστε κυρία Έλλης. Ευχαριστώ πολύ. Όταν ο Κόλιν Βέικφιλ και εγώ είχαμε την τιμή να προσφωνήσουμε την Επιτροπή πριν από έξι μήνες περίπου, εξηγήσαμε σχετικά με τη χωματερή τη θέση της ψηλά στην πόλη του Χότοντε Spring σε ασταθή πετρώματα με κατολισθήσεις από προηγούμενα ορυχεία κάρβουνο ε, είναι κοντά σε μαγαζιά και σπίτια, είναι πηγή ρήπανση για νερό και ατμόσφαιρα. Εξηγήσαμε ότι λείπει ε, κανονισμός ε, από τον αρμόδιο περιβαλλοντικό φορέα του Ηνωμένου Βασιλείου. Σημειώνουμε ότι ο οργανισμός αυτός του Ηνωμένου Βασιλείου απάντησε σε ερωτήσεις που ετέθησαν από την Επιτροπή αυτή και είναι κρίμα διότι δεν απάντησαν έντιμα και ειλικρινά. Τρεις παρατηρήσεις σε σχέση με την οσμή καταρχήν. Ε, οι στοχότων ε, υποφέρουν από την αποφορά. Καμιά φορά κρατάει μήνες από το 2000. Στον Ιούλιο φέτος ο οργανισμός ε, προσέφυγε στο δικαστήριο κατά της Μπίφα με βάση δύο από τις πολλές προσφυγές και καταγγελίες που είχε λάβει. Πρέπει να πούμε ότι η ε, είχε κάνει μήνυση στην πίφα κατά της οσμής ε, της αποφοράς αυτής και έκανε τη δουλειά της αλλά στην πραγματικότητα η φρικτή αυτή αποφορά είχε αναφερθεί πολλές φορές στον οργανισμό ε, και τους ζήτησαν να κάνουν έρευνα. Εκατοντάδες καταγγελίες. Ο ε, οργανισμός τις έστελνε στον, ε, υποτίθεται στον ε, διευθυντή της εταιρείας αλλά αυτός είπε ότι μόνο τρεις είχε λάβει. Επίσης είχε πει ότι δεν έχει σχέση με εμάς η αποφορά. Πολλές φορές μάλιστα ήταν προσβλητική και έλεγαν ότι το σπίτι της κυρίας που έκανε την καταγγελία μυρίζει. Επίση, ε, εμένα πολλέ φορέ ε, με είπε ότι με κατηγόρησε για κατασυρωή ψεύδη και ο οργανισμό πολλέ φορέ έγραφε ότι ερευνήθηκε και δεν είναι τεκμηριωμένε οι καταγγελίε ενώ δεν είχε γίνει έρευνα. Δεύτερον, για τα ύδατα και τη ρήπανση εκεί ε, αναφέρθηκε ότι υπήρχε ένας δρόμος για φορτηγά που είχε σταματήσει να υπάρχει τέλο πάντων και δεν υπήρχε από εκεί και πέρα ε, ρήπανση ενώ αυτό δεν είναι αλήθεια διότι υπάρχουν ε, αποπλήματα τα οποία έχουν διεισδύσει στα πετρώματα του υδροφόρου ορίζοντα και σε σημεία κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα ε, προϊόντα αυτά ε, έκκλησης, αποπλήματα ε, διείσδησαν και στην κυψέλη αυτή των επικίνδυνων αποβλήτων που είχαν μια επικάλυψη. Επίσης έχουν αναφερθεί ε, κάποια στοιχεία ε, απαντητικά που λένε ότι η πηγή της ρήπανσης ε, δεν είναι μεμονωμένο συμβάν αλλά υπάρχουν συγκεντρώσεις αμμονιούχου αζότου. Έτσι ε, αυτά είχαν γίνει ένα χρόνο πριν ε, δώσει στην Επιτροπή αυτή την εξήγηση σχετικά με το δρόμο τον παλιό για τα φορτηγά. Η ρήπανση των υδάτων έχουν αυξηθεί τώρα με το αμμονιούχο άζωτο και είναι 22,9 μιλιγκράμμ το λίτρο και όχι 16 μιλιγκράμμ το λίτρο που είπε η Επιτροπή στην, ε, οργανισμός στην Επιτροπή. Επίσης υπάρχουν στοιχεία που λέγουν ότι η μπίφα τώρα ζητάει τροποποιήσεις στην άδεια που έχει. Ε, ζήτησε στο Σεπτέμβριο του 2011. Ε, αυτές ε, οι τροποποιήσεις θα καταργούν πολλούς από τους ελέγχους συμπεριλαμβάνοντας τις, τα φρεάτια που, που έχουν ανοίξει επηρεάζουν τα όρια των αποπλημάτων, τα επίπεδα ε, και αυτό θα ισχύει για ακόμα 25 χρόνια και επίσης ε, μολυσμένες φαρμακευτικές ουσίες απόβλητα δηλαδή θα προσθεθούν στα 350 είδη αποβλήτων που υπάρχουν τώρα. Ε, αυτή δεν είναι μια αίτηση καθαρή και ειλικρινή. Εμεί έχουμε επίσης αντίγραφα ε, επιστολών που δείχνουν ότι ο περιβαλλοντικός οργανισμός συμφώνησε ήδη με τα αιτήματα της ΜΠΙΦΑ το Σεπτέμβριο του, και τον Οκτώβριο του 2010 και τον Μάρτιο του 2011. Και εκτό αυτού η ΜΠΙΦΑ πρόκειται τώρα να ανατινάξει εκατοντάδε κυβικών μέτρων των βράχων που περιβάλλουν τη χωματερή. Οι ρυθμιστικές αρχές ε, το επιτρέπουν αυτό ανεξάρτητα από την πολύ δυσμενή επίπτωση που θα έχει ε, στα πετρώματα γύρω-γύρω και στα σπίτια. Ε, πάλι οι πολίτες πρόκειται να ταλαιπωρηθούν. Οποιαδήποτε δράση λάβει ο περιβαλλοντικός οργανισμός θα είναι επιβλαβής ε, ήδη το απαγορευτικό κόστος σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στα δικαστήρια, η μπίφα μας κοροϊδεύει. Άλλη μια φορά ε, αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε σε αυτή την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προστασία, να μας προστατέψετε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Από την ε, Επιτροπή, αν θα ήθελε ε, κάποιος εκπρόσωπος να εκθέσει τη θέση, τη θέση της. Anybody from the... Ποιος θα μας πει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί, όπως ξέρετε, την αναφορά εδώ και αρκετό διάστημα και διερεύνησε πολλές ε, καταγγελίες. Πολλές είναι οι καταγγελίες βέβαια. Συνοψίζοντας, δεν θα επαναλάβω αυτά που ξέρει η Επιτροπή, η τελευταία μας ε, ανακοίνωση είναι του Σεπτεμβρίου. Προσθέτω μόνο ότι η θέση μας παραμένει. Ανησυχούμε γιατί ε, δεν ε, τακτοποιείται το θέμα και δεν διασφαλίζεται και η συλλογή των αερίων από εκεί. αυτό ήταν βασική προϋπόθεση. Αν η χωματερή διατηρεί το θα έπρεπε να μειώσει την ποσότητα υδάτων που εισέρχονται εκεί για να μειωθούν και τα αποπλήματα. Έτσι θα μειωθεί και η ε, αποφορά που ταλαιπωρεί τους κατοίκους. Αυτό που μας είπε αργότερα σε μετέπειτα ανακοίνωση τέλος Ιουλίου το Ηνωμένο Βασίλειο ε, είναι ότι η κάλυψη ε, έχει προχωρήσει και η συλλογή αερίων στη επίσης έχει προχωρήσει, αλλά θα πρέπει τώρα να τσεκάρουμε να δούμε τι άλλες δουλειές πρέπει να γίνουν. Παραμένει η ανησυχία. Δεύτερο ανησυχητικό θέμα το οποίο ετέθη πέρσι σε εμά είναι το θέμα της ρήπανσης των υπογείων υδάτων. Ε, Αυτά αυξημένα επίπεδα ρήπανσης στα υπόγεια υδάτα. Έτσι υπάρχουν ε, ενδείξεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο μας εξήγησε ότι αυτό ε, συνέβη ε, από ένα δρόμο ο οποίος τώρα δεν ε, λειτουργεί πια. Μας είπαν επίσης ότι σκέφτονται να κάνουν μήνυση κατά του, της επιχείρησης για αυτό το θέμα. Η Κομισιόν πρέπει να δει τώρα είναι στιγμιαίο το κακό, το, το αμάρτημα ή είναι κατά συρροή όπως λέει η αναφέρουσα και δείχνει ότι είναι πιο προβληματική και διαδεδομένη η ρήπανση. Ε, μετά από την αρχή της αναφοράς μας απασχόλησε να δούμε τι που έχει αυτή η κατάσταση στα υπόγεια ύδατα. Και ε, πριν ανοίξει η αναφορά, ε, ήδη υπήρχε φάκελος της Κομισιόν εδώ και το βασικό μέλημα και η ανησυχία ήταν αυτή, ε, ότι μπορούσαν να ε, χειροτερέψουν οι σχέσεις μεταξύ των ντόπιων και του οργανισμού περιβάλλοντος και να χαθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Γι' αυτό προβήκαμε στο ασυνήθιστο μάλλον βήμα να ζητήσουμε από ανεξάρτητο τρίτο να οριστεί για να εξετάσει την κατάσταση των υπογείων υδάτων στην περιοχή. Και συμφώνησαν οι Βρετανικές αρχές με την πρόταση αυτή όταν έκαναν την ε, έρευνα που ολοκληρώθηκε το 2006. Τώρα, η δυσκολία για την Κομισιόν είναι ότι είναι λίγο κινητό ο στόχο, θα λέγαμε, ε, ει ό,τι αφορά τη διαδικασία επί παραβάση, γιατί προφανώ θα πρέπει να, ε, η Κομισιόν να αποδείξει, να, να προσκομίσει αποδείξεις σε οποιαδήποτε δράση αναλάβει. Τώρα το πρώτο βήμα είναι να υποβληθεί ο, κατάλογο, ο φάκελος που ήδη υπήρχε για να αρχίσει η διαδικασία επί παραβάση ενδεχομένως Τώρα, με βάση τα νέα στοιχεία που πήραμε από την αναφέρουσα, θέλουμε άλλη μια φορά να επικοινωνήσουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο, να γίνει μια συνάντηση επί όλου του πακέτου και να δούμε πόσο προχώρησαν οι εργασίες κάλυψης, πώς προχώρησαν οι εργασίες συλλογή των αερίων και αυτό πολύ σημαντικό και ποια ήταν η έκβαση των ποινικών ε, ερευνών και άλλων ερευνών σε σχέση με την ενδεχόμενη επιδείνωση της ρήπανσης των υπογείων υδάτων στην περιοχή. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Καλά ακούγονται όλα αυτά και θα βοηθήσουν μάλλον. Αν και είναι κρίμα που χρειάστηκε 7 ε, χρόνια η αναφορά και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Επίσης δεν καταλαβαίνω Τι είναι το πρόστιμο αυτό των 27.000 λιρών στερλιτνών. Τι, ποιος θα αποζημιωθεί με αυτά τα λεφτά. Τέλος πάντων, ε, σίγουρα θα μείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και πιστεύω επίσης ε, και ο κύριος Τουρκάισε που έκανε έκθεση για τη διαχείριση αποβλήτων έχει καλύψει τα θέματά μας και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Υπάρχει και ε, περίπτωση να αποσταλεί επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου για να ενημερωθούμε περισσότερο σχετικά με το τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον, τι θα κάνουν σήμερα, τι θα κάνουν αύριο. Ευχαριστώ πολύ. for Mr. There is uh, number 16. Uh, Το 16. Το σημείο 16. σχεδιαζόμενες νέες εγκαταστάσεις χειμερινών αθλημάτων στο Μελάου και στο Ντάμουνς του Βοράλμπεργκ στην Αυστρία. Ίσως η Κομισιόν θα ήθελε να πει δύο λόγια για αυτή την αναφορά 672 στο νούμερο 16. Μπορείτε να μιλήσετε για το σημείο 16 Κομισιόν. Είμαστε δύο. Ε, εσείς αποφασίσετε, λέει η Πρόεδρος, ποιος θα μιλήσει. Okay. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, sorry for the delay, but... Ε, το συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ε, ακούσαμε μεγάλο ενδιαφέρον πάντων το ρουμανικό θέμα, τη ρουμανική αναφορά, γιατί συνδέεται με το σημείο που θα σας μιλήσω εγώ, που θα σας αναφέρω εγώ. Ευχαριστώ που δίνετε το λόγο στην Κομισιόν, που μας έδινε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την οδηγία περιβαλλοντικής επίπτωσης. Όπως είπατε, στην ετήσια έκθεσή σας για τις δραστηριότητε σας, αυτή η οδηγία περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι μία από τις οδηγίες που συζητιέται κάθε τόσο στις συζητήσεις της ε, Επιτροπής σας. Σε αυτή την περίπτωση εδώ έχουμε καλή, κακή εφαρμογή της εφαρμογής ε, της οδηγίας περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Αυστρία. Είναι κλασικό παράδειγμα οδηγίες, ε, της οδηγίας αυτής. Γιατί ε, συνδέεται με το πώς γίνεται η διαδικασία ε, εξέταση, screening. Η διαδικασία με βάση την οποία εξετάζουμε εάν ένα έργο θα πρέπει να υποστεί ε, μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου ή όχι. Υπάρχει ένα περιθώριο ευελιξία από πλευρά κράτου μέλου για να το αποφασίσει αυτό, είτε με τη δημιουργία κατοφλίων ή κάνοντα μία ανάλυση περίπτωση αναπερίπτωση. Είναι εντυπωσιακό αν δείτε τι στατιστικέ που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις περιπτώσεις αυτής της οδηγίας ε, και τις ε, ε, παραβάσεις που ξεκινάμε, οι 69% των περιπτώσεων παραβάσεων συνδέονται με αυτή τη διαδικασία του screening. Και από τις αποφάσεις του δικαστηρίου, το 80% συνδέονται με αυτό το πρόβλημα, δηλαδή προβληματικού, προβληματικής εξαίρεσης. Ο κύριος Βίλαντα ζήτησε από την Κομισιόν να απαντήσει σε δύο ερωτήσεις συγκεκριμένα. Πώς θα εγγυηθούμε ότι η εφαρμογή και η μεταφορά της οδηγίας αυτής θα γίνει σωστά σε όλα τα κράτη-μέλη και δεύτερον, αν πρέπει να τροποποιήσουμε την οδηγία ή τα παρατήματα για να εγγυηθούμε μια κοινή εφαρμογή αυτής της οδηγίας και των διατάξεών της. Θα προσπαθήσω καταρχά να σα περιγράψω τι μέσα έχει στη διάθεσή τη η Κομισιόν για να εξασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή και την ενιαία ε, ερμηνεία τη οδηγία στα κράτη-μέλη και, εν συνεχεία, θα αναφερθώ στην ε, διαδικασία επανεξέταση, αναθεώρηση τη οδηγία. Για να εξασφαλίσουμε ότι η οδηγία εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο και ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο στα κράτη-μέλη, κάνουμε μια συστηματική, ένα συστηματικό έλεγχο συμμόρφωσης. Εμείς αξιολογούμε δηλαδή πώς μεταφέρονται αυτές οι οδηγίες στα κράτη-μέλη και με βάση τις αναφορές και τα παράπονα που λαμβάνουμε αξιολογούμε τον τρόπο με τον οποίο η οδηγία εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Έχουμε και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από εθνικούς εμπειρογνώμονες από την, που ασχολούνται με την οδηγία αυτή για την περιβαλλοντική επίπτωση και συζητάμε εκεί ε, με τα κράτη-μέλη τις απόψεις μας για τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε ε, ενιαία την οδηγία. Ε, πέρα από, αυτά, από αυτές τις ομάδες που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε και στα κράτη-μέλη, στην Ισπανία και στην Ισπανία, ας πούμε, περιφερειακές και τοπικές αρχές συνεργάζονται ε, αρχές υπεύθυνες για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης, ετοιμάζουμε και ένα έγγραφο καθοδήγησης, όπου εξηγούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί η οδηγία και δίνουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουμε ένα έγγραφο καθοδήγησης για τη διαδικασία screening, πώς πρέπει να γίνει και πέρυσι δημοσιεύσαμε και ένα έγγραφο το οποίο αφορά την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Τέτοιου τύπου έγγραφα λοιπόν, τα οποία είναι στη διάθεση, στην ιστοσ... ε, διάθεσή σας στην ιστοσελίδα μας και έχουμε και άλλα έγγραφα, θα τα έχουμε έτοιμα μέχρι το τέλος του 2011, για την ε, οδηγία EIA και την ε, περιβαλλοντική αλλαγή και τη βιοπικιλότητα. Δηλαδή πώς θα αξιολογήσουμε ε, αυτά τα δύο στοιχεία, την κλιματική αλλαγή και τη βιοπικιλότητα στα πλαίσια της οδηγίας περιβαλλοντικών δικτώσεων. Επίσης, είχαμε τρεις συνεδριάσεις κατάρτισης με 80 περίπου δικαστές για να εξηγήσουμε, τους εξηγήσουμε τα προβλήματα με την οδηγία αυτή και παρά τις προσπάθειές μας έχουμε προβλήματα εφαρμογής στα κράτη-μέλη. Λογικό είναι στην περίπτωσή του screening γιατί κάθε χρόνο έχουμε 34.000 ε, προσπάθειες screening σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στατιστικά είναι αδύνατο λοιπόν κάποια στιγμή να μην προκύψει κάποιο πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα του screening δεν οφείλεται στο ότι διατάξει είναι ασαφή στην οδηγία. Η οδηγία όπως έχει συνταχθεί και όπως έχει εξηγηθεί και ερμηνευθεί από το δικαστήριο είναι σαφής, αλλά μερικές φορές τα προβλήματα εφαρμογής που αντιμετωπίζουμε οφείλονται στην έλλειψη πολιτικής θέλησης κάποιων αρχών, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε είναι περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να εφαρμόσουν σωστά την οδηγία. Μπορεί επίσης να μην έχουν και επαρκείς πόρους. Ε, άκουσα με ενδιαφέρον τη συζήτηση που κάνετε προηγουμένω. Γιατί όταν πρέπει να αξιολογήσουμε αν ένα ε, έργο ε, σέβεται την οδηγία αυτή, χρειάζεται κάποια πραγματογνωμοσύνη που μπορεί να μην την έχει το κράτο μέλο, ειδικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επίση, μπορεί να είναι πρόβλημα λόγω τη δομή δομής του, κράτους μέλους. Σε ομοσπονδιακά και περιφερειοποιημένα κράτη-μέλη έχουμε περισσότερα προβλήματα με την εφαρμογή της οδηγίας. Επομένως, λοιπόν, χρειάστηκε να διαρωτηθούμε μήπως πρέπει να αλλάξουμε την οδηγία, να την τροποποιήσουμε και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Και παρότι πιστεύουμε ότι είναι σωστή στη σύνταξή της, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα. Αλλά ακόμα και αν αλλάξουμε την οδηγία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτω ή άλλω ότι όλα θα εγγυηθούν. Γιατί όπω σα εξήγησα, ε, μπλέκονται πολλοί παράγοντε και φορεί αυτή τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, το 2009, με βάση μια έκθεση, ξεκινήσαμε μια δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση τη οδηγία περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου δηλαδή, και το αποτέλεσμα αυτή τη δημόσια διαβούλευση που έγινε το 2010 έδειξε ότι μία από τι βασικέ δυσκολίε είναι το screening γιατί δεν γίνεται συχνά με καλό τρόπο. Και έχει δύο επιπτώσει. Μερικέ φορέ κάποια έργα τα οποία θα έπρεπε να υπόκεινταν σε πλήρη μελέτη, γιατί έχουν σημαντικέ επιπτώσει, διαφεύγουν τη υποχρέωση. το άλλο πρόβλημα είναι ότι μερικέ φορέ τα κράτη-μέλη το παρακάνουν, δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο με την οδηγία και κάνουν τέτοιε μελέτε περιβαλλοντικού δικτύπου όταν δεν χρειάζεται. Ε, στα πλαίσια τη ε, αναθεώρηση, το πρόβλημα του screening, τη διαλογή των έργων, θα είναι από τα βασικά θέματα. Και η Κομισιόν θα προσπαθήσει να απλουστεύσει τη διαδικασία, να την κάνει πιο σαφής για το ποια έργα υπόκεινται και ποια δεν υπόκεινται, ούτω ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή. Αλλά ακόμα και αν την αλλάξουμε την οδηγία, το είπα προηγουμένω αυτό, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε 100% ότι θα εκλείψουν τα προβλήματα. Είναι αδύνατον η Κομισιόν να είναι δίπλα και να κρατάει το χέρι ε, σε κάθε αρχή, γιατί σας είπα ότι έχουμε κάθε χρόνο 34.000 τέτοιες διαδικασίες διαλογής. Αλλά και τροποποιώντας την οδηγίες και δίνοντας ενημέρωση και έτσι, κατευθυντήριες γραμμές, κατευθυντήριες αρχές, ε, νομίζω ότι θα εξασφαλίσουμε μια πιο ενιαία εφαρμογή της οδηγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να πω κάτι. γιατί είναι και θέμα του συνηγόρου των πολιτών. Πρέπει να ρωτήσουμε κάτι τους εκπροσώπους Επιτροπής. Η επιστολή του κυρίου Ποτότσνικ μετά την ερώτηση ξεκαθαρίζει ότι οι πίστες ΚΙ θα πρέπει να ε, στηρίζονται στην επιτυχή έκβαση της ΕΠΕ εξέταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Νομίζω ότι και η Κομισιόν εδώ φαίνεται να έχει τροποποιήσει λίγο την προσέγγιση της μέσα από αυτή την επιστολή, σε σχέση με αυτή την επιστολή. Γιατί ε, μέχρι τώρα οι εθνικές αρχές ήταν αρμόδιες για τις πίστες. Αν άλλαξε η άποψη της Κομισιόν, ερωτώ κι εγώ το θέμα ε, των χιονοδρομικών κέντρων πώς θα ρυθμίζεται νομοθετικά. Αυτή ήταν μια αναφορά, ε, μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλες και ίσως ε, είναι μια ευκαιρία για να ρυθμιστεί και να ξεκαθαρίσει το θέμα. Είναι και θέμα ανταγωνισμού, είναι και θέμα κόστους για αυτή την εγκατάσταση, το αν θα γίνεται μελέτη ΕΠΕ, αν θα υπάρχουν ε, περιβαλλοντικά ε, αντισταθμιστικά μέτρα κλπ. Όλα αυτά τα θέματα έχουν να κάνουν με πολλά λεφτά. Τα λεφτά αυτά και το κόστος θα πρέπει να ε, εν μέρη να ενσωματωθεί στις τιμές που θα αυξηθούν και δημιουργούνται πολλά και προβλήματα. Είπατε ότι τέλος του χρόνου θα υπάρξει νέα οδηγία. Θα έλεγα αυτή την αναφορά να την κρατήσουμε ανοιχτή μέχρι το Μάρτι και να δούμε πάλι αν η Κομισιόν τα guidelines τα έχει αντίστοιχα τροποποιήσει, τα έχει προσαρμόσει ή αν, καταλήξουμε, αν θα καταλήξουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει καινούργια οδηγία γιατί τα guidelines δεν θα είναι πια αρκετά, δεν θα επαρκούν. Με την αναφορά ανοιχτή, περιμένοντας το τελικό κείμενο... Α, ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Μια μικρή διευκρίνηση. Η πρόταση της Κομισιόν για την αναθεώρηση της οδηγίας θα είναι του χρόνου, στα μέσα του 2012. Τέλος του χρόνου θα προσθέσουμε καινούριο ε, έγγραφο για το guide, ε, guidelines για το περιβάλλον και την ΕΠΕ αλλά το πώς θα αξιολογούνται με βάση την ΕΠΕ, τα χιονοδρομικά κέντρα, ε, έχω ένα έγγραφο για το screening ήδη και υπάρχει και νομολογία του δικαστηρίου που λέει ξεκάθαρα ότι όταν τα κράτη-μέλη ε, είτε με ανάλυση κατά περίπτωση είτε με άλλο τρόπο δεν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μόνο το μέγεθος αλλά και τη θέση του κέντρου. Άρα λοιπόν δεν εξετάζουμε μόνο τον άμεσο αντίκτυπο αλλά και τον έμεσο αντίκτυπο των έργων. Αυτή η ενημέρωση παρουσιάζεται νομίζω ε, καλά στο τωρινό κείμενο των ε, guidance και σε σχέση με τις μελλοντικέ ΕΠΕ ένα στόχος θα είναι να ενσωματωθεί η νομολογία του δικαστηρίου στην ίδια την οδηγία για να είναι ε, σαφέστερη και να εφαρμόζεται με καλύτερο τρόπο. Ελπίζω να απάντησα στον αξιότιμο βουλευτή. Να κύριε ähm, Εντάξει, εντάξει. Θα ήθελα όμως μέχρι τότε το φάκελο να τον, να τον εξυγχρονίσουμε αν θέλετε ε, και στα πλαίσια της διερευνητικής αυτής ε, αποστολής. Επομένως κρατούμε την αναφορά ανοιχτή και τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πολύ. Uh, waiting. I'm informed that we are waiting. Ε, μου λένε ότι περιμένουμε τώρα τον συνήγορο του πολίτη ε, αν έχουμε ένα λεπτό. Είναι πραγματικά σκάνδαλο πώς αντιμετωπίζουμε το χρόνο των άλλων. Έχουμε τόσους αναφέροντες που θα πρέπει η γραμματεία να βρει άλλους χρόνους, να προβλέψει άλλους χρόνους. Ε, κανονικά ε, θα πρέπει να, πριν από μία ώρα να συζητηθεί το θέμα που με ενδιέφερε. Πέρασε μία ώρα. Πήγα αλλού και δεν ήξερα τι ώρα θα έρθει ο συνήγορο, ο διαμεσολαβητής. Πώς είναι δυνατόν να έρχονται από μια χώρα μέλος 20 και όλοι να θέλουν να μιλήσουν. Θα πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των αυτών που παίρνουν το λόγο αν δεν έχει δηλωθεί από πριν. Διότι θα πρέπει να δούμε και κάποια άλλα θέματα που αποτελούν και διεθνή αν θέλετε πολιτική. Κάνουμε υπόψη σας τις παρατηρήσεις σας. Να πούμε απλώς ότι η έλευση της διαμεσολαβήτριας ήταν έτσι κι αλλιώς για τις 11 η ώρα. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση που δεν ξέρω που οφείλεται, αλλά όχι στους ε, ε, καταγγέλλοντες ούτε στη διαδικασία θα το λύσουμε. Συμφωνώ με τον κύριο Βίλαντ. Ο χρόνος τρέχει και όταν ετοιμάζουμε την ημερήσια διάταξη εσωτερικά στην Επιτροπή να κάνουμε ε, μια κατανομή χρόνου που να την τηρούμε. Γιατί ο κύριος Βίλαντ είπε σήμερα ήρθα, ξανάρθα, έφυγα. Ε, η και επίσης και οι τελευταίοι αναφέροντες ζημιώνουν γιατί στην αρχή δίνουμε μπόλικο χρόνο και οι αναφορέ ε, στο τέλος και οι αναφέροντες που θα πρέπει να μιλήσουν στο τέλος τελειώνουν με συνοπτικές διαδικασίες. Θα πρέπει να λέμε ας πούμε πόσος χρόνος ε, ε, προβλέπεται γιατί είναι να διακόπτουμε γιατί είναι άδικο σε για τους τελευταίους αναφέροντες. Λοιπόν, χρειάζεται καλύτερος προγραμματισμός, ώστε κάθε αναφέρον που κάνει το ταξίδι στις Βρυξέλλες να έχει το δικαίωμα ίση μεταχείρισης και ίση ακρόασης, αν θέλετε. Θα αναφέρω, θα μεταφέρω τις παρατηρήσεις στη γραμματική. Θα το λύσουμε, κύριε Γιάρ να υποδεχτώ σήμερα την Πολωνή διαμεσολαβήτρια ε, και να ακούσουμε την εισήγησή της. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους σας και ευχαριστώ πάρα πολύ αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την πρόσκληση που μου έκανε και μου δίνει έτσι την ευκαιρία να έρθω και να σας παρουσιάσω την δουλειά του διαμεσολαβητή στην Πολωνία. έχουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Και αυτό ισχύει και για μένα, αλλά και για τους πέντε προκατόχους μου. Η θέση του διαμεσολαβητή κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα. Είναι κάτι πολύ θετικό. Αυτή είναι η εμπειρία μας, είναι πολύ θετική. Και όπως σας είπα, απορρέει από το ίδιο το Σύνταγμα. Η νομική βάση που έχουμε ε, μας οδηγεί σε διάφορες ε, διατάξεις και όπως σας είπα και στην αρχή οι πολίτες έχουν ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στον θεσμό του διαμεσολαβητή και όχι μόνο οι πολίτες αλλά και ξένοι ε, μετανάστες οι όσοι ζητούν άσυλο κτλ. Είναι θέμα του συντάγματος όπως σας το είπα Αναφέρεται εδώ τι ακριβώς λέει το Σύνταγμα στα αγγλικά, ότι δηλαδή ο διαμεσολαβητή πρέπει να φροντίζει να διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών σύμφωνα με τις διάφορε διατάξεις έτσι όπως αυτές ισχύουν. Το σημείο αυτό λοιπόν που αναφέρεται στο Σύνταγμα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν εξαρτάται από την εκάστοτε κυβέρνηση ή από την πολιτική κατεύθυνση της μίας ή της άλλης κυβέρνησης το θέμα εξάλλου των αποφάσεων του διαμεσολαβητή δεν έχει τεθεί ποτέ ε, σε αμφισβήτηση από καμία κυβέρνηση. Χρέος μας και καθήκον μας είναι να προστατεύουμε τα δικαιώματα των ατόμων, των πολιτών, που είναι κάτι διαφορετικό βέβαια από την δικαιοσύνη. Είναι διαφορετική δικιά μας δουλειά από εκείνη της δικαιοσύνης. Κάθε άτομο πρέπει να απευθύνεται και μπορεί να απευθύνεται στον διαμεσολαβητή στην Πολωνία και μπορεί να ζητήσει βοήθεια προκειμένου να υποστηρίξει τις ελευθερίες του, τα δικαιώματά του που πιστεύει ότι παραβιάζονται από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Οι πολίτες χρησιμοποιούν πολύ το δικαίωμα αυτό. Και βλέπουμε ότι έχουμε κάπου 50.000 προσφυγές οι οποίες απευθύνονται στον διαμεσολαβητή. Ο αριθμός αυτός εννοείται ότι αλλάζει κάθε χρόνο, πάντως είναι γύρω στις 50 με 65 χιλιάδες οι αιτήσει που φτάνουν σε εμά κάθε χρόνο. Πέρα λοιπόν από τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του διαμεσολαβητή της Πολωνίας υπάρχουν ε, και άλλα πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε. Έχουμε πολλές προσφυγές όπως σας είπα όλοι οι διαμεσολαβητές έχουμε να αντιμετωπίσουμε αντίστοιχα προβλήματα. Το συζητήσαμε αυτό μια φορά όλοι μαζί γιατί κάνουμε κατά καιρούς διασκέψεις. Πρόκειται βασικά για την παραβίαση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε για τον ιδιωτικό βίο είτε για τα οικονομικά δικαιώματα. Ο διαμεσολαβητής βέβαια δεν μπορεί πάντα να λύσει τέτοιου είδους παραβιάσεις. Αυτό που κάνω εγώ σε αυτή την περίπτωση είναι ότι απευθύνομαι στην υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή και μεταφέρω εκεί τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί υπάρχουν και άλλα ε, όργανα τα οποία μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση επιτόπου και να φροντίσουν και για αποζημίωση των ετούντων. Επιπλέον, βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται και άλλα μέσα που προσφέρει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε ο Πολωνός συνήγορος του πολίτη, ο διαμεσολαβητής, φροντίζει να χρησιμοποιήσει και αυτά τα μέσα. Είναι ένα θέμα που όλο και περισσότερο θα αντιμετωπίζουμε στο μέλλον. Στις περιπτώσεις αυτές, ο διαμεσολαβητής εξετάζει και βλέπει πώς αντέδρασαν οι αρμόδιες αρχές σε μία παραβίαση που έχει να κάνει με το αστικό δίκαιο ή με κάτι άλλο. Στη πρόσφατα υπήρξε μια τέτοια περίπτωση όπου εμείς παρεβήκαμε για να δούμε κατά πόσο η αστυνομία και οι τοπικές αρχές ε, που πήγανε σε κάποιο εστιατόριο αντέδρασαν με τον κατάλληλο τρόπο ή όχι και κατά πόσο οι κάτοικοι τη πόλη αυτή θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπίσει την υπόθεση αυτή διαφορετικά. Δηλαδή προσπαθούμε κάθε φορά να δούμε αν τηρούνται οι προδιαγραφέ έτσι όπως αυτές προβλέπονται ή όχι. Οι αρμοδιότητε μας στην Πολωνία επικεντρώνονται κυρίως σε παραβιάσεις που κάνουν οι εθνικές αρχές, σε τέτοιους ισχυρισμού. Δεν ασχολούμαστε δηλαδή με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η συνεργασία που έχουμε βέβαια με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή είναι μια εξαίρετη συνεργασία. Και θέλω να πω εδώ στην Επιτροπή σας και να μιλήσω για ένα σχέδιο το οποίο ελπίζω πολύ σύντομα να προχωρήσει βάσει των επαφών που έχουμε. Τι θέλουμε. Θέλουμε όλοι οι διαμεσολαβητές στην Ευρώπη να έχουν ένα ενιαίο αριθμό τηλεφώνου. Αυτό θέλουμε, αυτό ελπίζουμε. Όπως έχουμε το 112 που είναι για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, έτσι το ίδιο να ισχύει και για τους διαμεσολαβητές ολόκληρη την Ευρώπη. Ταξιδεύουμε, μερικές φορές, πολλές φορές ε, θα έλεγα, ότι διαπιστώνουμε πως οι πολίτες μας, οι οποίοι μετακινούνται πολύ, ε, διαπιστώνουν παραβίωση των δικαιωμάτων τους και μερικές φορές αναγκάζονται να χάσουν πάρα πολύ χρόνο και χρήμα για να καταλάβουν πώς μπορούν να φτάσουν, να έχουν πρόσβαση στον διαμεσολαβητή της χώρας του. Ενώ αν υπήρχε ένας ενιαίος αριθμό τηλεφώνου, τον οποίο να το γνωρίζουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να μπορούν να επικοινωνήσουν με του διαμεσολαβητέ του. Υπάρχει η Διεθνή επίση οργάνωση και θα έπρεπε εύκολα να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε. Είναι κάτι που στην πράξη μπορεί να βοηθήσει πολύ. Οι πολίτε έτσι σιγά σιγά θα μάθουν καλύτερα τα δικαιώματά του και θα μπορούν πιο εύκολα να τα υποστηρίξουν. Αυτό είναι ισχύει για όλου του Ευρωπαίου πολίτε και για όλου όσου ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πιο συγκεκριμένα για την Πολωνία πάλι. Εμεί εξετάζουμε το θέμα των ελευθεριών, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά επίσης μας απασχολεί πολύ και το θέμα της ίσης μεταχείρισης των ατόμων. Είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ από 1η Ιανουαρίου. Γιατί, γιατί προσπαθήσαμε όλη αυτή τη χρονιά να ετοιμάσουμε ό,τι οι δομές χρειάζονται για τη στήριξη των δικαιωμάτων αυτών. Βέβαια, δεν είχαμε όλα τα οικονομικά μέσα που θέλαμε, δυστυχώς, αλλά ελπίζω, ελπίζω ότι σιγά σιγά θα καταφέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα με τον επόμενο προπολογισμό. Χάρη όμως στη συνεργασία μας με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, επίσης με οργανώσεις ειδικών, μπορέσαμε να δημιουργήσουμε τρεις επιτροπές εμπειρογνωμόνων για θέματα ε, διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων, των μεταναστών και των ατόμων με αναπηρίες. Κάθε μία από τις τρεις αυτές επιτροπές ειδικών δούλεψε και προχώρησε σε διάφορες δράσεις. Υπάρχει επίσης και μία κοινωνική ομάδα η οποία βοηθάει στις δράσεις αυτές στα πλαίσια των διακρίσεων. Έτσι λοιπόν μπορώ να σας πω εδώ ότι τα μέσα ενημέρωσης και η κοινή γνώμη φρόντισαν να προωθηθεί μια δράση με συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίας στις επόμενες εκλογές, την Κυριακή όπως ξέρετε έχουμε. Θα είναι η πρώτη ευκαιρία όπου θα έχουμε μια τόσο μεγάλη δράση στην οποία συμμετέχουν οι διάφορες τοπικές επιτροπές εκλογών ώστε να δούμε τελικά ποιο είναι ο καλύτερος χώρο μέσα στον οποίο μπορούν να λάβουν χώρα εκλογές αυτές, ώστε και τα άτομα με αναπηρία που είναι 2 εκατομμύρια στην Πολωνία να μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές απρόσκοπτα. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που μπορώ να σας πω ότι με τη συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα. Ολόκληρη η κοινωνία συμμετείχε και ο ίδιος ο πρόεδρος, ή το γραφείο του Προέδρου συμμετείχε επίση στη δράση αυτή για να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στι εκλογέ. Για την ίση μεταχείριση πρέπει επίσης να έχετε υπόψη σας ότι είναι ένα διακυβερνητικό θέμα. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης γι' αυτό, οπότε εγώ το μόνο που κάνω είναι ότι ελέγχω και ερευνώ. Και γι' αυτό ενημερώνομαι για το τι δομές διαθέτουμε και πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις έτσι όπως αυτές προβλέπονται. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να ξέρετε ότι αναλαμβάνει διάφορες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες. Κάθε φορά που βλέπουμε ότι υπάρχει μια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων ενός πολίτη, είτε μας έρχεται από έναν ιδιότητα, είτε μας έρχεται από μια οργάνωση, είτε από μια περιφέρεια, ή για παράδειγμα από τον διαμεσολαβητή για τα δικαιώματα του παιδιού. Κάθε φορά εμείς αντιδράμε και εξετάζουμε πώς έχει η κατάσταση από την αρχή. Υπάρχει πάντως μεγάλη αύξηση των προσφυγών που μας φτάνουν, όπως βλέπετε και σε αυτό το, σε είτε πρόκειται για προσφυγές από ιδιώτες είτε από οργανώσεις. Από το 2000 μέχρι το 2010 βλέπετε εδώ την εξέλιξη. Και αυτό που βλέπουμε το 2010, η τελευταία στήλη δηλαδή που υπάρχει μια μείωση, έχει να κάνει με τον τραγικό θάνατο του ε, δόκτωρα και του προκατόχου μου. Είναι βέβαια κάτι πολύ προσωπικό το ότι έχασε τη ζωή του ότι ο προηγούμενος ε, πέρασαν πάρα πολλοί μήνες μέχρι να ξαναρχίσει η δουλειά μου, μέχρι να αναλάβω εγώ και να ε, προχωρήσουμε με τις προσφυγές. Έχουμε 255 προσωπικό. Να ξέρετε ότι όλοι ε, ταυτίζουν, ταυτίζονται προσωπικά με τον διαμεσολαβητή. Και έτσι λοιπόν υπήρξε αυτή η τραγική εξέλιξη το 2010. Τώρα το 2011 σίγουρα θα φτάσουμε στα επίπεδα όχι μόνο του 2009, αλλά θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι προσφυγές. Θέλω να υπογραμμίσω επίσης, κυρίες και κύριοι, ότι ο ρόλος του διαμεσολαβητή στην Πολωνία έχει να κάνει κατά πολύ με το γεγονός ότι οι αιτήσει που έρχονται δεν είναι δεν, έχουν, δεν πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη μορφή ούτε κοστίζουν. Απλώς πρέπει να υπάρχει μια υπογραφή. Το γεγονός ότι έχουμε τόσες πολλές προσφυγές και γίνονται δωρεάν είναι επειδή μπορούν να γίνουν και μέσω του διαδικτύου. Και προφορικά μάλιστα και μερικές φορές προφορικά υποβάλλουν τις αιτήσει τους οι άνθρωποι. Είναι ένας τρόπος αυτός για να αντιμετωπίζουμε ε, θέματα τα οποία δεν είναι πολύ αναπτυγμένα νομοθετικά στην Πολωνία. Οι δράσεις μας επιτόπου ε, γίνονται σε συνεργασία και με τους δικαστικούς συμβούλους. Και πολλές φορές τα θέματα αυτά λύνονται επιτόπου. Δεν λέω ότι θέλουμε οπωσδήποτε να δώσουμε τη δουλειά μας σε άλλους, αλλά πάντως με τη συνεργασία μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα. Κάποιος μπορεί να έρθει στο γραφείο μας, να δει τις πρακτικές που ακολουθούμε κάθε φορά που έχουμε μια προσφυγή από ένα πολίτη. Γίνονται συνομιλίες, για παράδειγμα, και με τους αναφέροντες. Πρέπει να ξέρετε πίσω το 2010, τι περιπτώσεις ε, υποβλήθηκαν στην υπηρεσία του διαμεσολαβητή. Η δομή και η διάρθρωση αυτή επαναλαμβάνεται σε όλους τους διαμεσολαβητές λίγο πολύ. Υπάρχουν και κάποια νέα θέματα, αλλά υπάρχουν ίδιοι και τα ίδια θέματα που έρχονται και επανέρχονται, γιατί το θεωρούν πολύ σημαντικό οι πολίτες. Το γεγονός ότι εδώ βλέπετε κάποια, κάποιες μικρές περιπτώσεις για ορισμένα θέματα. Πρόκειται για τις απαντήσεις που δώσαμε μέχρι τώρα για να ολοκληρωθεί μια υπόθεση. Και υπάρχουν και πολλές νέες περιπτώσεις όπως σας είπα. Εδώ βλέπετε τις νέες περιπτώσεις. Και βλέπετε επίσης πως τον πρώτο χρόνο είχαμε πάρα πολλά θέματα. Ό,τι είχε προκύψει κατά την κομμουνιστική περίοδο, ξαφνικά εκείνη τη χρονιά ε, ήρθαν ως προσφυγές προς τον ε, διαμεσολαβητή. Μετά υπήρξε μια σχετική μείωση. Αλλά βλέπετε ότι μετά υπήρξαν και νέες περιπτώσεις, ξανά και ξανά, που έπρεπε να αναλυθούν σοβαρά και σε βάθος. Πώς γίνονται τώρα οι διερευνήσεις. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον διαμεσολαβητή. Να ξέρει κατά πόσο μπορεί να δεχτεί, να θεωρηθεί παραδεκτή δηλαδή μια προσφυγή και μετά πώς θα ενημερώσει τον αναφέροντα για το τι σκοπεύει να κάνει. Έπειτα απευθυνόμαστε στις αρμόδιες αρχές, εκτός αν αποφασίσουμε να αρνηθούμε ως μη παραδεκτή την προσφυγή. Πάντως 60% περίπου των αιτήσεων που μας φτάνουν γίνονται παραδεκτές. 4% ε, συνήθως πρόκειται για μια νομική υπηρεσία. Δηλαδή λέμε στους ε, ετούντες ότι πρέπει να απευθυνθούν σε μια άλλη υπηρεσία για να λύσουν το θέμα τους. Αυτό το θέμα της ε, πληροφόρησης έρχεται ως βοήθεια και πολλές φορές από τους βουλευτές ή από τους βοηθούς τους γιατί συχνά οι αναφέροντες πριν φτάσουν σε εμά έχουν απευθυνθεί σε κάποιο βουλευτή. Έτσι και οι γερουσιαστές και οι βουλευτές βοηθάνε. Πολλές ε, βέβαια περιπτώσεις δεν προχωρούν και τα προβλήματα είναι πολλά. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το θέμα του ποινικού δικαίου. Ο διαμεσολαβητής Ε, χρησιμοποιείται σε βάση OPCAP. Οι πολίτες μάλλον ενημερώνονται από τις δικαστικές αρχές πολλές φορές για το ότι πρέπει να απευθυνθούν στον διαμεσολαβητή. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα, όπως είναι θέματα δημόσιας διοίκησης, υγείας, δικαιωμάτων ε, των ξένων. Είχαμε πολλές εξελίξεις πάντως και σε μία σειρά θεμάτων που είχαν να κάνουν με παραβιάσεις από τα μέσα ενημέρωσης. Πολλές παρεμβάσεις υπήρξαν και καταλήξαμε τελικά σε θετικά συμπεράσματα για τους πολίτες, σε θετικές καταλήξεις, για παράδειγμα για μια οικογένεια Μογγόλων. Φέτος πάντως προσπαθήσαμε πολύ περισσότερο να λύσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις και να βελτιώσουμε την διαδικασία. Στο λίγο χρόνο που έχω εγώ στη θέση μου, ο πρόεδρος Κομαρόσκι υπέγραψε ένα νόμο βάσει του οποίου θα έχουμε νέες περιπτώσεις που θα μπορεί να επεξεργαστεί ο διαμεσολαβητής. το θέμα του, της νομοθεσίας αυτής, κατάργησης, είναι ένα θέμα το οποίο θα προχωρήσει και θα βοηθήσει πολλούς. Αυτό που προσπαθεί να πετύχει η νομοθεσία είναι να υπάρχουν τα μέσα που χρειάζονται για αρκετούς μήνες. Ο Πολωνός Διαμεσολαβητής έχει διάφορες αρμοδιότητες. Τις βλέπετε εδώ. Μπορεί να πάει επί τόπου, να εξετάσει από κοντά ένα θέμα να έχει επαφή με τη δικαιοσύνη, με το δικαστικό σώμα και μπορεί να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη κάθε φορά που το κρίνει χρήσιμο για να ζητήσει επεξηγήσεις ή πληροφορίες. Στην Πολωνία πιστεύουμε ότι ο διαμεσολαβητής έχει τεράστιες αρμοδιότητες και μερικές φορές αυτό οδηγεί σε προβλήματα με την ποινική διαδικασία. Γιατί εμείς μπορούμε να παρεύουμε μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί μια δικαστική διαδικασία. Αλλιώς δεν μπορούμε να παρέμβουμε, πρέπει να περιμένουμε και μας χρειάζεται χρόνος. Μερικές φορές μπορεί να υπάρξει στραβιδίκηση, να υπάρχει λάθος και εμείς καλούμεθα να βρούμε το λάθος και να βρούμε και τη λύση. Υπάρχουν διάφορες ε, διατάξεις που αναφέρονται στο έργο του διαμεσολαβητή. Εδώ ε, βλέπετε ότι κάνουμε και εμείς ε, κάτι σαν και αυτό που κάνετε και εσείς εδώ στην Επιτροπή Αναφορών σας. Δηλαδή έχουμε διάφορες αναφορές που εξετάζουμε που έχουν να κάνουν με διαδικασίες πειθαρχικές για παράδειγμα Και θα μπορούσε επίσης να είναι κάτι αυτό που βοηθάει και στην εκπόνηση της νομοθεσίας, παρόλο που εμείς δεν έχουμε νομοθετική αρμοδιότητα και ούτε λέω ότι τη θέλουμε. Με τίποτα δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά εμείς συνεργαζόμαστε με τους βουλευτές, όπως σας είπα, κάθε φορά που πιστεύουμε ότι αυτό χρειάζεται. Εδώ βλέπετε ποιες είναι οι γενικές αναφορές που μας φτάνουν πέρυσι, δηλαδή το 2010. Βλέπετε ποιες είναι οι κύριες ε, αναφορές. Είναι πολλά και διαφορετικά θέματα. Ένα νέο στοιχείο πάντως, κατά τη διάρκεια της δικιάς μου θητείας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικές φορές δεν ξέρω ο πού να απευθυνθεί, η καινοτομία λοιπόν είναι κάποιε συνεδριάσεις στι οποίε συμμετέχει και ο υπουργό Δικαιοσύνη και άλλοι υπουργοί από την κυβέρνηση. Σε μια τέτοια συνάντηση αυτό που γίνεται είναι ότι εγώ τους ενημερώνω, του πληροφορώ και του εξηγώ πώ θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία ή τους λέω ποια είναι τα θέματα των δικών του δικήσεων, των δικών του υπουργείων που δεν λειτουργούν ικανοποιητικά και οδηγούν σε αναφορέ τέτοιες συναντήσεις ήταν πολύ χρήσιμες γιατί είδαμε ότι οδήγησαν σε αλλαγές κυρίως στην πολωνική δικαιοσύνη. Εδώ τώρα μπορείτε να δείτε στη διαφάνεια αυτή ποιοι απευθύνουν ε, υποθέσεις επίσης σε εμάς. Βλέπετε ότι είναι το δικαστήριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, ε, Υγείας κλπ. Και εδώ βλέπετε ποιες είναι οι αρμοδιότητες του διαμεσολαβητή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρεμβαίνει όταν διαπιστώνεται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Και το συνταγματικό δικαστήριο και το ανώτατο δικαστήριο και το διοικητικό. Πέρυσι εγώ απευθύνθηκα σε όλα αυτά τα όργανα για το στεγματικό Δικαστήριο ο διαμεσολαβητής μπορεί να προχωρήσει σε διάφορες ε, διαδικασίες. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να φροντίσει για τη συμμετοχή σε διάφορους τομείς που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Δεν λέω ότι έχουμε πολλές προσφυγές, αλλά έχουμε πάντως αρκετές που μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι. Ο προκάτοχός μου απευθύνθηκε στο συνταγματικό δικαστήριο όταν επρόκειτο για την διάκριση σε βάρος των ηλικιωμένων ατόμων. Είχε να κάνει το θέμα με το δικαίωμα στη συνταξιοδότηση, έτσι ώστε να έχουν δικαίωμα σε σύνταξη ηλικιωμένοι. Ήταν κάτι που δουλέψαμε πολύ στην προηγούμενη θητεία του διαμεσολαβητή. Το βλέπουμε σε διάφορα επαγγέλματα. Οι συμβολιογράφοι, για παράδειγμα, ή για τους εκπαιδευτικού υπήρχε πρόβλημα με τις συντάξεις των ηλικιωμένων. Δεν λέω ότι τα λύσαμε όλα. Στην περίπτωση των συμβολιογράφων ε, μπόρεσα να λύσω κάποια προβλήματα. Εδώ τώρα με τους ε, εκπαιδευτικούς ήταν αλλιώ, γιατί και εγώ ήμουν πριν εκπαιδευτικός και μου είναι δύσκολο να ασχοληθώ με ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το ίδιο το δικό μου το συμφέρον. Το Συνταγματικό Δικαστήριο πάντως αντιμετώπισε τις αιτήσει που έφταναν από τον διαμεσολαβητή. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Βλέπετε τι αιτήσει έχουν υποβληθεί στο συνταγματικό δικαστήριο και ποιες είναι οι διαδικασίες όσον αφορά προσφυγές από πλευράς της δικιάς μου υπηρεσίας. Αν μη τι άλλο γίνεται συζήτηση για τέτοια θέματα, ακόμα και αν δεν δοθεί λύση άμεσα με τους συνεργάτες μου μερικές φορές βλέπω ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε στο σταγματικό δικαστήριο. Αν μη τι άλλο όμως διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κάποια αλλαγή στην οτροπία, ότι το συζητιέται αυτό το θέμα στο σταγματικό δικαστήριο, μπορεί να υπάρξει μια οργάνωση που να υποβάλει προσφυγές στη συνέχεια ώστε να αλλάξουν τα πράγματα, να υπάρξει κάποια αλλαγή αν μη τι άλλο. και εσείς τη γνωρίζετε αυτή τη διαδικασία, γιατί αυτό ακριβώς θέλετε και εσείς να κάνετε η κοινωνία να ενημερωθεί και να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τα θέματα τα οποία εξετάζετε κι εσείς. Οι αποφάσεις πάντως του Συνταγματικού Δικαστηρίου για τις δικές μας τις προσφυγές ε, διαπιστώνουν που υπάρχει το ασύμβατο με το Σύνταγμα. Στο ανώτατο δικαστήριο της Πολωνίας εκεί φτάνουν άλλα θέματα. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν έχουν προετοιμαστεί πάντα καλά οι προσφυγές αυτές. Είτε δεν έχουμε ακολουθήσει την σωστή διαδικασία, οι πολίτες δηλαδή προηγουμένως για να φτάσουν εκεί, ενώ ξέρουμε ότι το ανώτατο αυτό δικαστήριο είναι το ανώτατο ακριβώς όργανο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί κανείς. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα στο έργο μου. Είναι δράσεις με τις οποίες ασχολούμαι αυτή την εποχή. Αν δω ότι στο πρώτο στάδιο δεν υπάρχουν αποτελέσματα, στη συνέχεια προσπαθώ να οργανώσω μία δημόσια συζήτηση για το θέμα χ ότι πρόκειται για την ασφάλεια των άστεγων, για παράδειγμα. Μετά από τη δημόσια συζήτηση, κάνω μία δημόσια δήλωση. Απευθύνομαι στο Υπουργείο Δικαιοσύνη, διοικητικέ αρχέ και αν δω ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή από εκεί, μια που υπάρχουν διάφορες απόψεις, δεν συμφωνούν πάντα όλες οι αρχές για το πώς καταγράφονται οι συνομιλίες μας για παράδειγμα, αυτό που γίνεται είναι ότι πάμε στο συνταγματικό δικαστήριο. Αλλά αν μη τι άλλο, εφόσον έχει προηγηθεί δημόσια συζήτηση και εφόσον έχει γίνει δήλωση από τη δικιά μου την πλευρά, η κοινή γνώμη, αν μη τι άλλο, κατανοεί καλύτερα τις παραμέτρους του κάθε θέματος. Δεν είναι δηλαδή συζήτηση αυτή μόνο για τους ειδικού, αλλά και για την κοινή γνώμη, για τον κόσμο. Και όταν το θέμα είναι πολύ ειδικό, τότε οργανώνουμε δημόσια συζήτηση, ακόμα και μια ε, διάσκεψη με ερευνητέ. Είναι κάτι που κάναμε, για παράδειγμα, όταν επρόκειτο για την προστασία του ιδιωτικού βίου και των ε, ατομικών δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι και κυρία Πρόεδρε άλλη μια φορά για την πρόσκλησή σας. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι πέρα από τις αρμοδιότητες που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν αλλαγές, ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια πολύ. Και γιατί? Γιατί υπήρξε πίεση από την κοινωνία των πολιτών σε πολλές περιπτώσεις. Οι δημόσιες αρχές πιστεύαν ότι ε, ο διαμεσολαβητής τι θα είναι, εντάξει ας τον αφήσουμε να δουλέψει και αυτός, θα βοηθήσει λιγάκι. Έτσι θα είναι και απόδειξη ότι έχουμε ελεύθερε εκλογές, ε, κοινοβούλιο κτλ. Γι' αυτό δώσανε αρμοδιότητε στο διαμεσολαβητή. Μετά όμω η κοινωνία των πολιτών άλλαξε, απίτησε ακόμα περισσότερε αρμοδιότητε, και αυτό διαπιστώνουμε ότι όλο και περισσότερε αρμοδιότητε έχει ο διαμεσολαβητή στην Πολωνία. Αυτά είχα να πω. Κυρίες και κύριοι, περιμένω τις ερωτήσεις σας τώρα. Είμαι στη διάθεσή σας για να έχουμε μια καλή συζήτηση. Εγώ να ευχαριστήσω την Πολωνή διαμεσολαβήτρια, την καθηγήτρια κυρία Ιρένα Λίποβιτς. Ε, η διαδικασία λέει, όπως μου λένε στη, από τη Γραμματεία, ότι μπορούμε να απευθύνουμε γενικής φύσεως ερωτήσεις ε, στην κυρία Λίποβιτς ε, και στη συνέχεια θα παρακολουθήσει μαζί μας τις αναφορές τριών από τρεις Πολωνούς ε, ε, Ευρωπαίους πολίτες ε, επομένως η πρωινή συνεδρία θα κλείσει με την παρουσία της ε, κυρίας Λίποβιτς και τους ε, καταγγέλλοντες από την Πολωνία. Αν υπάρχουν ερωτήσεις γενικές που να αφορούν στην εισήγηση της κυρίας Λίποβιτς. Ναι κύριε äh, äh, Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν κυρία Λίποβιτς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας Ευχαριστώ και για τον συνάδελφο Βαλέσα, ο οποίος είχε ένα ατύχημα και του ευχόμεθα καλή ανάρρωση για να έρθει γρήγορα στην Επιτροπή μας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εμείς παλεύουμε στην ίδια γραμμή με το που εσείς ως διαμέσολαβητής, εμείς ως Επιτροπή Αναφορών τασόμεθα υπέρ των συμφερόντων των πολιτών, είμαστε υπεύθυνοι για αυτά. Είμαστε ένα σεισμογράφος του λαού, αν θέλετε, ως ένα βαθμό, γιατί και σε μας και σε εσά απευθύνονται άμεσα οι πολίτε χωρίς φίλτρα, χωρίς ε, διοικητικού διαμεσολαβητές και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Η Επιτροπή Αναφορών και ο διαμεσολαβητής είναι δείγματα μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Και το λειτουργήμά σας πραγματικά είναι απαραίτητο. Έξι ερωτήσεις έχω. Με κοιτάει αυστηρά η πρόεδρος, γιατί πρέπει να τηρηθεί και ο χρόνος βέβαια, το ξέρω. Μου κάνει εντύπωση η ποικιλία των υποθέσεων που καταπιάνεστε. Απλοϊκό ερώτημα από την πλευρά μου. Πόσο μεγάλη είναι η ομάδα των συνεργατών σας, πόσους ε, απασχολείτε στο γραφείο σας και στην ομάδα, μας, ε, σας. Δεύτερον, μπορείτε να μας πείτε κάτι για τη μέση διάρκεια διοικητικής ας πούμε, διεκπαιρέωσης. Πόσο γρήγορα θα απαντηθεί η ερώτηση του πολίτη ή θα δοθεί συνέχεια στην καταγγελία του. Τρίτον, βάζετε κι εσείς κάποια όρια και λέτε ε, ας αν μέχρι τότε δεν λυθεί το πρόβλημα θα πρέπει ειλικρινώς να ομολογήσω στον πολίτη ότι δεν μπορώ να σε βοηθήσω αλλά θα πάρεις μια απάντηση. Τέταρτη ερώτηση, κάτι πολύ ενδιαφέρον για μένα. Ελπίζω να κατάλαβα καλά. Εσείς δηλαδή μπορείτε να κάνετε άμεσα έρευνες απευθεία. Δηλαδή, μάθατε κάτι από τα μέσα ενημέρωση ότι κάποιο ε, αντιμετωπίστηκε άσχημα. Εκεί μπορείτε εσεί να κάνετε έρευνα, μπορείτε επίση να προσφεύγετε απευθεία, γιατί είπατε ότι μπορείτε και στο δικαστήριο, αν θέλετε, να είστε διάδικο, Μπορείτε να μας τα εξηγήσετε, γιατί εγώ ε, καινούρια τα ακούω όλα αυτά. Πέμπτη ερώτηση. Είπατε ότι μπορείτε να ε, καταργείτε δικαστικές αποφάσεις. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Πώς γίνεται δηλαδή. Δηλαδή όταν αποφαίνεται ένα δικαστήριο και αποφασίζει μπορείτε εσείς ας πούμε να ανατρέψετε τις δικαστικές αποφάσεις. Τέλος, μαζί με την Επιτροπή Αναφορών στο Πολωνικό Κοινοβούλιο, αν υπάρχει τέτοια, υπάρχει Επιτροπή Αναφορών στο Πολωνικό Κοινοβούλιο και αν υπάρχει, πώς συνεργάζεστε με την Επιτροπή αυτή. Και πάλι ευχαριστώ που ήρθατε και που μας μιλήσατε. Ε, just a moment. Thank you very much for your many... Ευχαριστώ πολύ για τις πολλές ερωτήσεις σας που αντιφάσκουν σε αυτό που είπατε πιο πριν για το χρόνο, αλλά εγώ το τηρώ. Ο, ο κύριος Μποστινάρου πρώτα. Όχι ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία γενική παρατήρηση θα κάνω μόνο. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά, αλλά δεν εκπλήσωμαι. Που βλέπω πόσο μεγάλο ρόλο και πόσες εξουσίες έχετε και στον τομέα της αλλαγής του δικαιικού συστήματος αν χρειάζεται και πώς κάνετε ε, νομική προσφυγή αν επιβάλλετε, πόσες αρμοδιότητες έχετε σε θεσμικό επίπεδο για να δράτε και να αντιδράτε μαζί με άλλες αρχές στην Πολωνία. Μπορεί το πολωνικό παράδειγμα να αποτελέσει υπόδειγμα και για κάποιους άλλους εθνικούς διαμεσολαβητές όταν καλούνται να προασπίσουν τα δικαιώματα των πολιτών γιατί δεν συμβαίνει πάντα αυτό να παίζουν τόσο ορατό ρόλο. Ε, και μια ερώτηση μόνο κυρία Λίποβιτσε ποιες είναι οι σχέσεις σας με το Πολωνικό Κοινοβούλιο, δηλαδή θεσμικά πώς εργάζεστε και τι αντίκτυπο έχει ε, το δικό σας έργο όταν πάτε σε μια επιτροπή του Κοινοβουλίου, δηλαδή τι αντίκτυπο έχει στο έργο του Κοινοβουλίου η παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι συντομότατος. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσίαση και ζητώ συγγνώμη που έπρεπε να φύγω για λίγο για να δεχτώ μια κλίση. Και εγώ εντυπωσιάζομαι με τις δράσεις αυτές. Ίσως ξέρετε ότι σήμερα το πρωί εξετάζαμε πάλι μια αναφορά κατά των πολωνικών αρχών που αρνούνται να δώσουν ένα πιστοποιητικό ληξιαρχική ερωτικής πράξης ε, για κάποιον αν είναι παντρεμένος ή διαζευγμένος. Πρόκειται για ζευγάρια που θέλουν να έρθουν σε ένωση δύο φίλου ε, πρόσωπα σε μια άλλη χώρα. Οι πολωνικές αρχές παλιότερα είχαν πει ότι είναι συνιστά διάκριση αυτή η άρνηση. Εσείς μιλάτε για την ε, προάσπιση ελευθεριών όταν περιορίζονται, θα διαφυλάσω μελέτε τις ελευθερίες, είστε υπέρ της αρχής της ίσης μεταχείρισης, της δίκαιης μεταχείρισης δεν συμφωνείτε ότι δεν είναι δίκαιη η μεταχείριση αυτή και θα εξετάσετε την υπόθεση αυτή για λογαριασμό των Πολωνών ε, πολιτών που είναι 50 και στους οποίους αρνούνται να χορηγήσουν αυτό το πιστοποιητικό ληξιαρχικής πράξης αν είναι ε, ανήπαντροι ή ε, παντρεμένοι. Δεν πρόκειται για ένωση που θα λάβει χώρα στην Πολωνία, αλλά σε άλλη χώρα, εκτός πολωνικού εδάφους, σε ένα από τα άλλα 16 κράτη-μέλη που εγκρίνουν και νομιμοποιούν τις ενώσεις ατόμων ιδίου φύλου. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Ε, μπορεί ε, η κυρία Λιποβίτς να απαντήσει. Ε, ε, ε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάρ, για τις εξαιρετικές ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Εις ό,τι αφορά τον αριθμό όχι το, του προσωπικού, έχουμε 265 που εργάζονται στο γραφείο μας είναι αρκετός ο αριθμός. 250 νομικοί μπορούν να μας βοηθήσουν να μελετήσουμε τις τρέχουσες υποθέσεις. Φέτος ε, έχουμε αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες στον τομέα της ίσης μεταχείρισης και χρειάστηκε να απασχολήσω με 15 άτομα για να καλύψουμε τις άμεσες ανάγκες. Μέχρι τώρα πάντως χειριστήκαμε επαρκώς τις υποθέσεις που είχαμε με αυτούς τους 250-265 ε, συνεργάτες. Τώρα για τα χρονικά μας περιθώρια ε, χειρισμού μιας υπόθεσης. Διαφέρει. Καμιά φορά η απάντηση δίνεται σε λίγες μέρες μέσα αν όμως πρέπει να περιμένουμε ε, κάποια νομικές διευκρινήσεις, μπορεί να περάσουν και 4-3-5 πέντε μηνες μέχρι να συμπληρωθούν τα στοιχεία στο νομικό φάκελο. Μπορεί τα στοιχεία να πάρουν μήνες μέχρι να μας έρθουν. Και ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι πολλές φορές παίρνει χρόνο ο χειρισμός τέτοιων περίπλοκων ε, υποθέσεων και φακέλων. Καμιά φορά ε, ολοκληρώνουμε 10 υποθέσεις την ημέρα όταν είναι απλή νομική απάντηση. Αν είναι περίπλοκο το θέμα, ή αν ε, ε, εισέρχεται και η απόφαση δικαστηρίου, παίρνει μήνες υποθέσεις. Κατά μέσον όρο πάντως μια απλή περίπτωση ολοκληρώνεται σε ένα μήνα και όταν είναι πιο σύνθετη η υπόθεση όπου θα πρέπει δηλαδή να ζητήσουμε φακέλους ε, από το δικαστήριο, εκεί μπορεί να μας πάρει και 6-7 μήνες. Τώρα για την ενεργό παρέμβαση σε διαδικασίες Για το φόρτο εργασίας μας πρέπει να πω ότι έχουμε κάποια προβλήματα οικονομικά και στις υποθέσεις της ΑΠΚΑΤ είχαμε προβλήματα χειρισμού πολλές φορές. Τώρα για τις δικαστικές αποφάσεις μπορούμε να ζητήσουμε να ακυρωθεί μια δικαστική απόφαση σε περίπτωση αμέλειας ή ε, νομικών σωλμάτων. Αυτό είναι ένα δικαίωμα ενός διαδίκου σε μια υπόθεση. Ο διαμεσολαβητής όμως επίσης μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού. και έχω 30 μέρες στη διάθεσή μου για να ε, ζητήσω ακύρωση δικαστικής απόφασης. Καμιά φορά μπορούμε να ζητήσουμε ακύρωση αν ένας διάδικος σε μια υπόθεση δεν μπόρεσε να ζητήσει την ακύρωση για οποιονδήποτε λόγο σε περίπτωση ας πούμε ε, έκδοσης προσφύγων αν αποφασίσω ότι οι πολωνικές αρχές έχουν παραβιάσει το δίκαιο, την νομοθεσία, τότε υποστηρίζω τον πρόσφυγα και τον, ή την βοηθώ στην υπόθεση του της. Αν βέβαια κάποιοι πληρεξούσιοι ε, υποστηρίξουν τον διάδικο στη δικαστική, στην εκδίκαση της υπόθεσης πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε κάτι τέτοιο γιατί με αυτόν τον τρόπο αποστέλουμε συγκεκριμένο μήνυμα στην ευρεία κοινή γνώμη. Οι 260 άνθρωποι βέβαια που εργάζονται σε μας δεν αρκούν για να συμμετέχουν σε εκατοντάδες δικαστικές υποθέσεις. Αυτή λοιπόν η διαδικασία γίνεται κατ' εξαίρεση. Αλλά έχει τύχει να, ε, κάνω, να ε, χειριστώ υποθέσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας και με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αυτά τα ε, συμβάντα ρατσισμού ή άδικης αντιμετώπισης της μειονότητας των Ρώμα τότε στέλνω αντιπροσώπους για να ε, εποπτεύσουν ή να παρακολουθήσουν την ε, εκδίκαση της υπόθεσης. Είναι σημαντικές υποθέσεις αυτές. Θα ήθελα να πω ότι εργαζόμεθα πάρα πολύ καλά με την ε, Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου, του Bundestag, του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Και οι συνάδελφοί μου συμμετέχουν σε διάφορες συναντήσεις γερμανικών φορέων και οργανισμών. Είναι πολύ καλό αυτό το παράδειγμα της συνεργασίας μας. Και χάρη στην πολωνογερμανική συνεργασία άρχισε ένα πρόγραμμα το οποίο μας επιτρέπει να προστατεύουμε ανθρώπους που μεταναστεύουν στη Γερμανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο και γίνονται και είναι άστιγοι. Έχουμε ένα πρόγραμμα και με το προξενείο της Πολωνίας στο Αμβούργο που βοηθάει αυτούς τους αστέγους. Συχνά πρόκειται για ανθρώπους που τους έχουν ξεγελάσει οι ενδιάμεσοι, οι μεσάζοντες. Κάποιους έπρεπε να τους ξαναστείλουμε στην Πολωνία. Η συνεργασία αυτή μεταξύ Πολωνίας-Γερμανίας σε αυτό το τομέα είναι πολύ καλή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μποστινάρου για τα σχόλιά του και να υπογραμμίσω ότι οι συναντήσεις μας με την Επιτροπή Αναφορών και άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου αυτού είναι σε τακτά διαστήματα, είναι πολύ τακτικές Οπότε πράγματι έχουμε τακτικές επαφές με κοινοβουλευτικά σώματα. Δεν μπορώ όμως να συμμετάσχω στην παρασκευή νομοσχεδίων στο Πολωνικό Κοινοβούλιο, γιατί αν το έκανα αυτό τότε δεν θα μπορούσα να διαμαρτύρομαι και να φέρνω αντιρρήσεις αν υπάρξει πρόβλημα σε κάποιο νομοσχέδιο ή νόμο. Μπορώ να γνωμοδοτώ χωρίς να συμμετέχω όμως στην εργασία σχεδιασμού της νομοθεσίας. Δεν μπορώ να παρασκευάζω νομοθεσία και να την ελέγχω ταυτόχρονα, δεν γίνεται αυτό, είναι ασυμβίβαστα αυτά. Επίσης έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε ε, να λάβουμε το λόγο ενώπιον του Πολωνικού Κοινοβουλίου για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επί παραδείγματι. Και αυτό το δικαίωμα, ε, δεν, ε, αυτού του δικαιώματος δεν κάνουμε χρήση υπερβολικά. Κατά την έναρξη της θητείας του, ο διαμεσολαβητής εκφωνεί λόγο στο Πολωνικό Κοινοβούλιο και μπορεί να ε, λάβει το λόγο οποτεδήποτε το επιθυμεί αργότερα. Να προσθέσω επίσης ότι ε, έχουμε κοινοβουλευτική συνεργασία και με άλλα κοινοβούλια όπως το Bundestag και προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε πολλές ε, ε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συνεργαζόμεθα και με την αρμόδια επιτροπή γι' αυτό της Γερουσίας. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Κάσμαν. Θα ήθελα να πω ότι για το συγκεκριμένο ερώτημα αυτό αφορά τις αναφορές που θα εξετάσουμε, είναι αναφορές από την Πολωνία, τις οποίες τις έχουμε μελετήσει όλες. Εν προκειμένου, στην υπόθεση που αναφέρει, αναφέρεται, στην οποία αναφέρεται ο κύριος Κάσμαν, εγώ προσέφυγα στις πολωνικές αρχές για να καταργηθούν οι αδίποτε εμπόδια, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της χορήγησης ή ασδήποτε άδεια. Εγώ στις 15 Μαρτίου προσέφυγα στις πολωνικές αρχές με το αίτημά μου και έλαβα απάντηση από τον Υπουργό Εσωτερικών. Ο Υπουργός απάντησε θετικά στην παρέμβασή μου και συμμερίζεται την άποψή μου ότι αυτά τα θέματα πρέπει να λυθούν. Αντιλαμβάνουμε λοιπόν ότι η υπόθεση του κυρίου Μπίντρον θετικά επελήθη. Θα φροντίσω τώρα η απάντηση και η υπόσχεση του Υπουργού των Εσωτερικών να τεθεί σε εφαρμογή, να πραγματοποιηθεί. Ο νέος Υπουργός μετά τις εκλογές θα ε, φροντίσω να σεβαστεί την υπόσχεση που έδωσε ο προκάτοχός του. Έχω όμως επίσημη επιστολή από τον Υπουργό των Εσωτερικών και φαίνεται ότι το ζήτημα λύθηκε. I would also like to express my... Και εγώ να εκφράσω την έκπληξή μου, θετική έκπληξη, για τις εξουσίες αυτές που σας δίνει το πολωνικό δίκαιο σε εσά την ε, Πολωνή διαμεσολαβήτρια. Νομίζω ότι η κυρία Λίποβιτς θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τους ομόλογους της μέσω του Ευρωπαίου Ομπούτσμαν μέσω του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και να κάνει μια συζήτηση για να τους εξηγήσει τις αρμοδιότητές τη. Πάρτε αυτή την πρωτοβουλία και εμείς σα υποστηρίξουμε. Μικρόφωνο. αντιστρέψαμε τη σειρά των αναφορών. Υπάρχουν δύο αναφορές ακόμα. Η μία από τις αναφέρουσες ήρθε ειδικά από το Βερολίνο για να μιλήσει. Δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή της και ελπίζω να λυθεί το πρόβλημα, να μπορέσει να μιλήσει δηλαδή. Δύο μέρες έχει μόνο στη διάθεσή της. Η πρόεδρος μιλάει. Εντυπωσιάζομαι επίσης από το βαθμό συμμετοχής των πολιτών στις εργασίες σας. Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ζητήσω να δώσετε προσοχή σε, ένα, σε μια πολύ επικίνδυνη τάση που αναδύεται στην Ευρώπη. Κάνουμε λόγο συνέχεια για σχέδια λιτότητας. Ορισμένες κυβερνήσεις τα χρησιμοποιούν ως πρόσχημα για να ξεφορτωθούν τα γραφεία περιφερειακών διαμεσολαβητών ε, Φερρυπίν, αυτό συμβαίνει στην Ισπανία ή στην Ιταλία. Φυσικά είναι θέμα των εθνικών κυβερνήσεων αυτό, είναι θέμα κρατών μελών. Ε, ειδικά σε εποχές λιτότητας, οι διακρίσεις μπορεί να αυξηθούν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορέσουν οι διαμεσολαβητές να συνεισφέρουν ε, σε μια μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα στην Ήπειρό μας. Ε, θα ήθελα σκεφτείτε λίγο αυτό το πράγμα. Το θέτω προς ε, ενημέρωση και προβληματισμό σας. Δεν θα το ξεχάσουμε. Να συνεχίσουμε τώρα με το σημείο 20. Κυρία Ενρίκα Γκλέν, Γκλέντς.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 οι Πολωνοί που διαμένουν στο εξωτερικό δεν μπορούν να λάβουν τα έγγραφά τους. Πρόκειται για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ε, πλήττονται συνήθως, δεν μπορούν να παραστούν καν στις, ε, στην εκδίκαση των υποθέσεων γιατί απλώς δεν έχουν λάβει τα έγγραφα. Ε, γιατί δεν μπορούν οι πολωνικές αρχές να προσθέσουν μια διάταξη ούτως στο σχετικό νομοσχέδιο, ούτως ώστε να σεβαστούμε τον κανονισμό 1393 του 2007 για την επίδοση των δικαστικών εγγράφων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για όλους τους Πολωνού, τους Πολωνούς που διαμένουν εκτός Πολωνίας ανά την Ευρώπη. Να σας μιλήσω για μια άλλη περίπτωση, ε, μια αναφορά που συνδέεται πάρα πολύ με την ε, αναφορά που μόλις ακούσατε. Και οι δύο αναφορές αφορούν τα προβλήματα επίδοσης των εξοδίκων και δικαστικών εγγράφων στην Πολωνία. Ο πολωνικός νόμος, η πολωνική νομοθεσία δεν ε, λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στην κοινωνία, δηλαδή οι άνθρωποι μετακινούνται, ζουν σε άλλα κράτη από, αυτά, από τα οποία γεννήθηκαν και η κοινωνία πρέπει να προσαρμόζεται. Η, αναφέρω, η αναφέρουσα που έγραψε την επόμενη αναφορά, 277 κάθετος 2010, μου ζήτησε να διαβάσω μια δήλωση. Τι διαβάζω. Είναι δύσκολο να, να φανταστούμε μια πραγματική ολοκλήρωση και τα πλεονεκτήματα αυτή τη ολοκλήρωση, ό,τι αφορά πούμε, την ελεύθερη κυκλοφορία, εάν είναι αδύνατον οι Ευρωπαίοι πολίτε να ανταλλάσσουν επιστολέ ελεύθερα ούτε μεταξύ τους, ούτε μεταξύ αυτών και των θεσμικών οργάνων. Ε, μιλάω για έγγραφα τα οποία αφορούν δικαστικές υποθέσεις. Περί αυτού μιλάει η αναφορά η δική μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει μια ειδική ανακοίνωση που μας την έστειλε και την έστειλε στους ευρωβουλευτές και που μιλάει για θέματα δικαστικά, αλλά και όχι μόνο. Μιλάει κυρίως για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πάνω απ' όλα και για την ε, σωστή και επαρκή επίδοση των εγγράφων των δικαστικών υποθέσεων, αλλά και των εξοδίκων πράξεων. Θέλουμε να υπάρχουν κάποιες κοινέ διαδικασίες για ποινικά θέματα, για διοικητικά θέματα, για δικαστικές υποθέσεις, για εξοδικαστικές υποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση που μας έστειλε μιλάει για διακρίσεις εναντίον κάποιων πολιτών λόγω εθνικότητας. Οι αναφέροντες λένε ότι το θέμα δεν είναι θέμα διάκρισης λόγω εθνικότητας, είναι διάκριση μάλλον λόγω κατοικίας, λόγω του ότι κάποιος διαμένει σε ένα άλλο κράτος μέλος από αυτό το οποίο γεννήθηκε. Αυτά είναι από τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελευθερία κυκλοφορίας. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη στην απάντησή της τα όσα είπα. Συνοψίζοντας, πρέπει να αποδείξουμε ότι η Πολωνία... Πρέπει να πούμε μάλλον ότι η Πολωνία με την εσωτερική νομοθεσία της μέχρι στιγμής αγνοεί το ευρωπαϊκό δίκαιο στις διοικητικές διαδικασίες οι Πολωνοί πάλι στέλνουν τα έγγραφα διαταχυδρομείου. Όμως το Μάιο του 2011 αλλάξανε ρότα. Λάβαμε πληροφορίες από τα λεγόμενα επαρχιακά γραφεία στην Πολωνία ότι Τώρα άλλαξαν τα πράγματα και ένας νομικός, νόμιμος εκπρόσωπος ή αντίκλητος πρέπει να προσδιοριστεί από τον Πολωνοπολίτη. Δεν στέλνουν δηλαδή, τα έγγραφα στο εξωτερικό, αλλά θέλουν να ξέρουν ποιος είναι ο αντίκλητος του Πολωνού που διαμένει στο εξωτερικό, ο οποίος θα λάβει ε, μία επιστολή. Αλλά αυτό σε, σε εποχές ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι επιπλέον εμπόδιο. Αντί να καταρρύπτουμε τα εμπόδια, δημιουργούμε νέα δηλαδή. Αν θέλουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα νομοθετήματά μας είναι τέτοια, ούτως ώστε να διευκολύνουν όλους όσους διαμένουν σε διαφορετικά μέλή να τους βοηθούν σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή επιστολών. Είτε αυτά αφορούν ποινικά θέματα, διοικητικά θέματα, είτε εξοδικαστικά θέματα εν γέννη. Και οι δύο αναφορές τελικά δηλαδή αναφέρονται στο ίδιο πρόβλημα, στην επίδοση των δικαστικών εγγράφων. Επαναλαμβάνω. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κινείται προς μία κατεύθυνση, αλλά εμείς και εμείς τρέχουμε κατά πόδας. Δεν ε, υπάρχει μια διαφορά φάσης και ως εκ τούτου υπάρχουν πολλά εμπόδια τα οποία κανονικά πρέπει να καταρριφθούν. Mr. and Mrs. Kranovska uh, uh, will, say the positions of the committee. Of the... Τώρα οι δύο εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεχεία η Δημεσολαβήτρια από την Πολωνία. Σε ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Είναι ίδιες οι αναφορέ ω προς το θέμα τους. Θα απαντήσω ε, σε θέματα που αφορούν αστικές υποθέσεις και συνάδελφος ε, σε θέματα που αφορούν ποινικές υποθέσεις. Για την επίδοση ε, γράφων σε διοικητικές υποθέσεις, δεν υπάρχει ενωσιακό μέσο. Το άρθρο 1 του κανονισμού 1393 ε, του 2007 για την επίδοση των εγγράφων λέει ότι ο κανονισμός δεν ισχύει σε διοικητικά θέματα, σε διοικητικές υποθέσεις. Σε acta jure imperi δεν έχουμε δηλαδή μέσο, δεν έχουμε εργαλεία, δεν έχουμε νομοθέτημα στα χέρια μας για διοικητικές υποθέσεις. Όμως, Ε, Όμω, σε σχέση με το άρθρο 1135 του Πολωνικού Κώδικα, η Κομισιόν πιστεύει ότι το άρθρο αυτό παραβιάζει το κανονισμό για την επίδοση των δικαστικών εγγράφων. Στις 17 Μαρτίου του 2011 η Κομισιόν ήρθε σε επαφή με τις πολωνικές αρχές και έλαβε δύο μήνες μετά μία απάντηση από το, Υπουργείο, από το Δικαιοσύνης Πολωνίας που είπε ότι είναι έτοιμο να αλλάξει τις διατάξεις αλλά η απάντηση ήταν αρκετά σαφής. η Κομισιόν ετοίμασε, ετοίμασε μια επίσημη επιστολή που θα σταλεί σύντομα στις πολωνικές αρχές ως ανταπάντηση. Ο άλλος εκπρόσωπος της Επιτροπής θα απαντήσω εν συντομία για τα ποινικά θέματα. Η συντάκτρια της αναφοράς, μιλάω για τη δεύτερη, όχι, διορθώνει τώρα, για την πρώτη αναφέρουσα λέει ότι το άρθρο 5.1 για την δικαστική αλλοβοήθεια σε ποινικέ υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης του 2000 για τον, την επίδοση των δικαστικών εγγράφων που λέει ότι η άμεση ή η ταχυδρομική επίδοση των εγγράφων σε άτομα που διαμένουν α, σε ένα άλλο κρατός μέλος δεν εφαρμόζεται από τα πολωνικά δικαστήρια. Μιλάω για τα ποινικά πολωνικά δικαστήρια. Η συντάκτρια λοιπόν της αναφοράς ισχυρίζεται ότι ο νομοθέτης έχει επιβάλει κανονισμούς περιοριστικούς Λέει μάλλον ότι μπορεί να επιδοθούν και με ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα έγγραφα. Θα μπορούσαν να επιδοθούν με αυτούς τους δύο τρόπους. Το θέμα είναι η Κομισιόν μπορεί να νομοθετήσει αυτόν τον τομέα. Εδώ και λίγο καιρό από τη συνθήκη της Λισαβόνας μπορούμε να παρέμβουμε για τη δημιουργία κοινών ελάχιστων κανόνων σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων. Αναφέρω ένα κατάλογο που αναφέρει στο άρθρο 82 η συνθήκη. Μιλάμε για τους ελάχιστους κανόνες σε ό,τι αφορά το παραδεκτό των, αποδείξεων, το, τα δικαιώματα των θυμάτων και τα δικαιώματα των προσώπων στις ε, ποινικέ υποθέσεις. Η επιλογή όμως του νομοθέτη και δεν είναι απεριόριστη. Περιοριζόμαστε από αυτό το άρθρο, το οποίο αναφέρει κάποιους τομείς και έχουμε και κάποιες ε, πολιτικές προτεραιότητες αλλά και νομικές. Υπενθυμίζω τον οδικό χάρτη που υιοθέτησε το 2009 το Συμβούλιο το οποίο θέλει να ενισχύσει τα δικονομικά δικαιώματα των ε, υπόπτων, των ε, διοκόμων, διο, κατα, κατηγορούμενων σε ποινικέ υποθέσεις και θα πρέπει να παρουσιάσουμε κάποιε πρωτοβουλίες σταδιακά σε πολύ συγκεκριμένους τομείς. Εδώ αναφέρομαι στις εργασίες που έχουν ξεκινήσει, την οδηγία για τη μετάφραση των εγγράφων, την οδηγία για πρόσβαση σε δικηγόρο, την οδηγία για τα δικαιώματα του κατηγορουμένου κτλ. Μιλάω, για, εδώ, μιλάω τώρα για τομείς προτεραιότητας. Όχι, διορθώνει η ομιλήτρια. Πρόκειται για βασικά δικαιώματα. Νομίζω όμως ότι το θέμα της άμεσης ε, αποστολής των εγγράφων δεν εντάσσεται σε αυτόν τον κατάλογο. Τώρα, αν η Κομισιόν μπορεί να διώξει το κράτος μέλος γιατί δεν σέβεται τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση για την Δικαστική Αλληλοβοήθεια, Διαπιστώσαμε ότι ο κώδικας ποινική δικονομία προβλέπει στην περίπτωση όπου ο διάδικος διαμένει σε ένα άλλο κρατός μέλος ότι τα πολωνικά δικαστήρια προσφεύγουν στην επίδοση εγγράφων μέσω αντικλήτων ή μέσω ε, αντιπροσώπου του και μετά ζητούν από την δικαστική αρχή της άλλης χώρας να επιδώσει τα έγγραφα. τώρα, είναι περίπλοκη όντω αυτή η διασυνοριακή επίδοση, γιατί ο πολωνικός κώδικας υποχρεώνει του τους Πολωνούς που διαμένουν σε ένα άλλο κρατός μέλλον να κοινοποιήσουν την ταχυδρομική διεύθυνση του υπεύθυνου στην Πολωνία. Μια ταχυδρομική διεύθυνση δηλαδή στην Πολωνία. Επομένως, τα έγγραφα τελικά δεν επιδιώνται κατευθείαν σε αυτούς. Υπάρχουν λοιπόν ε, κάποιες ε, ελλείψεις εδώ. Έχετε κάποια λύση. Ναι, ναι, θα έρθω σε αυτό το θέμα. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Αλλά σας υπενθυμίζω το πλαίσιο. Εδώ μιλάμε για μια σύμβαση. Από το παλιό καθεστώς που δεν εφαρμόζεται όμως άμεσα και έχουμε τη δυνατότητα από το 2014 στην αλλά δεν ακούμε. Μιλάτε και οι δύο μαζί. Προς το παρόν δεν υπάρχει λύση. Γιατί αυτά τα μέτρα δεν είναι μέτρα προτεραιότητας, δεν είναι προτεραιότητά μας. Και δεν μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να διώξουμε το κρατό μέλο. Ευχαριστούμε πολύ που μας ενημερώνετε για τι δυνατότητε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ήρθα στην ε, συνεδρίασή σα, παρόλο που δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Αναφορών. Πήρα αυτή την ελευθερία γιατί πριν από μερικού μήνες έστειλα μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό μετά από αίτημα των ετούντων και πήρα μια απάντηση πολύ παρόμοια με αυτή που μόλις ακούσαμε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δείχνει ότι υπάρχει διάκριση όταν πρόκειται για την επίδοση δικαστικών ε, ή εξοδικαστικών ε, εγγράφων. Όταν πρόκειται για τα διοικητικά δεν έχουν να μας πούνε. Αλλά όταν πρόκειται πάντως για ε, διαδικασίες ποινικέ που χρειαζόμαστε περισσότερες εγγυήσεις, που πρόκειται για τα δικαιώματα όλων των διαδίκων, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπορούμε με τον ίδιο τρόπο να παίρνουμε τα έγγραφα όπως και όταν πρόκειται για αστικές, εξοδικαστικές και διοικητικές διαδικασίες. Πρόκειται για περιπτώσεις που δεν είναι τόσο ευαίσθητες όπως είναι οι ποινικέ, οπότε γιατί όχι. Ρωτάω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν βλέπετε εσείς διάκριση να υπάρχει ε, όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση όταν υπάρχουν ξεκάθαρα εμπόδια στην περίπτωση επίδοσης ε, και εξοδικαστικών ε, εγγράφων. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει κάποια στιγμή η Επιτροπή. Εμείς κρατούμε την ε, καταγγελία ανοιχτή και φροντίζουμε να βρούμε λύση στο ερώτημα. Να προχωρήσουμε στην επόμενη, επειδή ο χρόνος ε, μας κυνηγάει. Mm-hmm. Ε, ε, could you answer to all of them? Could you answer to all of them at the end? Μπορείτε να απαντήσετε στο τέλος σε όλες, γιατί περιμένει και ο αναφέρον. Είναι αναφορά πάλι από την Πολωνία που έχει να κάνει... Can I say something? Oh yes, κύριε. Ja Χαίρομαι που είναι εδώ και διασαμιλαβητής. Έτσι κι αλλιώς η Επιτροπή θα πρέπει κάποια στιγμή να μας απαντήσει. Θα περιμένουμε την απάντηση και ελπίζω να έχουμε κάποια απόφαση. Λοιπόν, χαίρομαι που είναι μαζί μας η διαμεσολαβήτρια, διότι όταν είναι κανείς σε αυτή την αίθουσα, καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι και πόσο προβληματικό είναι ακόμα και σε αυτό το στάδιο, πόσο μάλλον στη συνέχεια. Το βλέπετε με τέτοια σας τα μάτια ότι με την πολωνική νομοθεσία δημιουργούνται προβλήματα. Το βλέπετε τώρα, χαίρομαι γι' αυτό. Και ελπίζω εσείς και η ομάδα σας να ξεκινήσετε να πάρετε κάποια βήματα δηλαδή για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Γιατί όπως βλέπετε κάποιες διαδικασίες στην Πολωνία δυστυχώ, δεν είναι σωστέ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σα έχουμε μαζί μα σήμερα. Ε, να ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής αυτής ε, εκ μέρους της εκστρατείας καμπάνια Πρέτσκιου Ομοφίβη, θέλω που είναι εκστρατεία κατά τη ομοφοβία. Θέλω να σα ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε για άλλη μια φορά την αναφορά μα. αναφέρον ε, αναφέρεται σε διαδικασίε τη Πολωνία που αρνούνται να χορηγήσουν πιστοποιητικό οικογενειακή κατάσταση... σε Πολωνούς πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να συνάψουν σχέση καταχωρημένη συμβίωση ή γάμο με άτομο του ίδιου φίλου σε άλλο κράτο μέλο. Από τότε που η Πολωνία έγινε μέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλοί γκέις και λεσβείς από την Πολωνία επιθύμησαν να συνάψουν γάμους ή να έχουν μία μόνιμη σχέση με άτομο του ίδιου φίλου. Βέβαια σε χώρες εκτός της ε, άλλες χώρες, όχι μέσα στην Πολωνία, αλλά σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, προπόθεση για να καταχωρηθεί τέτοιο πιστοποιητικό είναι να πρόκειται για άτομα διαφορετικού φύλου. Δυστυχώς η πολωνική δίκηση ενέκρινε μια πολιτική η οποία αρνείται τέτοια πιστοποιητικά λοιπόν σε ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι επιθυμούν να συνάψουν γάμο με άτομα του ίδιου φίλου εκτός της Πολωνίας. Συγχρόνως οι πολωνοί πολίτες περιμένουν Ε, που πρόκειται να συνάψουν γάμα με άτομο διαφορετικού φύλου εκτός Πολωνίας δεν έχουν κανένα πρόβλημα για να πάρουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Η οργάνωσή μας λοιπόν έχει πάρει πάνω από 50 ε, διαμαρτυρίες, καταγγελίες από Πολωνούς πολίτες, ε, ομοφιλόφιλους ή λεσβίες που σκοπεύουν να συνάψουν γάμο εκτός Πολωνίας. Οι ίδιοι δημόσιοι υπάλληλοι αναγνωρίζουν ότι απορρίπτουν πολύ περισσότερες τέτοιες αιτήσει στις ε, διάφορες πόλεις και τα χωριά της Πολωνίας. Βασιζόμενοι σε προδιαγραφές που ισχύουν στην Πολωνία για ε, τις περιπτώσεις των ομοφιλόφίλων. Πρόκειται λοιπόν για μία διάκριση. Η δικιά μας η οργάνωση υποστηρίζεται από την διαμεσολαβήτρια μια που πρόκειται για διαδικασίες διακρίσεων. Πρόκειται για τα παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η νομοθεσία της Πολωνίας παραβιάζει τον οικογενειακό βίο και τον ιδιωτικό βίο των πολιτών αυτών. Και μόνο το όνομα που ζητάνε του ατόμου με το οποίο σκοπεύει αυτός που ζητάει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να συνάψει γάμο και μόνο το ότι ζητάνε το όνομα αυτό δείχνει ότι πρόκειται για άτομο του ίδιου φίλου και έτσι είναι αδύνατον να πάρουν τα πιστοποιητικά αυτά. Δεν έχουν υπάρξει τροποποίησεις μέχρι τώρα στην υπάρχουσα νομοθεσία. Δεδομένη της ε, εντολή που έχει δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέλει οι θεμελιώδει ελευθερίες να τηρούνται από τα κράτη-μέλη και δεδομένου της διακριτική ε, φύσης της πολιτικής ενός κράτους μέλους που παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία, ζητούμε από τα ευρωπαϊκά κοινοτικά όργανα να αναλάβουν δράση για να διορθωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εγώ ευχαριστώ για τη συντομία σας. Ε, ας έχουμε δύο παρεμβάσει παρεμβάσεις από τον κύριο Κάσμαν. Πρώτα από την Commission. First the Commission. Yes, please. Uh... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς πρέπει και εγώ να πάω πάρα πολύ γρήγορα γιατί έχει προχωρήσει η ώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν γνωρίζει την κατάσταση αυτή στην Πολωνία εδώ και καιρό. Και σας είπαμε και την προηγούμενη φορά που ήρθαμε εδώ ότι θα αναλάβουμε δράση και το κάναμε. Στείλαμε επιστολή λοιπόν από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη στις Πολωνικές Αρχές το Μάιο όπου λέμε ότι η άρνηση αυτή για το οικογενειακό πιστοποιητικό μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας και κατοικίας των πολιτών εκείνων οι οποίοι θέλουν να συνάψουν γάμο ή μόνιμη, συμφωνία σε άλλη χώρα εκτός Πολωνίας με άλλον πολίτη. Πήραμε λοιπόν ε, απάντηση και με υποφελούμε από την ευκαιρία που είναι εδώ η Πολωνή Διαμεσολαβήτρια για να σας πω ότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποια κίνηση όσον αφορά τις πολωνικές αρχές από τα τέλη Αυγούστου με την επιστολή αυτή που μας στείλαν. Όμως η ε, απάντηση αυτή δεν είναι συγκεκριμένη, δεν αναφέρεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για δράσεις που θα αναλάβει προκειμένου να αλλάξει τρέχουσα πρακτική. Οπότε διαρθρώνεται σε δύο τμήματα και θέλω να σας ενημερώσω για αυτά. Πρώτον, έχουμε το τμήμα όπου αιτιολογεί, αιτιολογούν οι πολυνικές αρχές ε, το θέμα της αντίδρασής τους και γιατί αρνούνται το πιστοποιητικό αυτό και λένε οι πολωνικές αρχές ότι θα συνεχίσουν την πρακτική ελέγχου των προϋποθέσεων κατά πόσο δηλαδή μπορεί να συνάψει γάμο ή όχι σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία το άτομο το οποίο ζητάει το ε, πιστοποιητικό αυτό κατάστασης. Και εκεί έρχομαι τώρα στο δεύτερο τμήμα, αναφέρεται ότι συζήτηση, γιατί έτσι λένε, συζήτηση αναφέρεται στα πολωνικά, έτσι μεταφράζεται στα αγγλικά, discussion, ότι ξεκίνησε η συζήτηση προκειμένου να πάψει η ρύθμιση αυτή. Κάτι το οποίο συνάδει και με αυτά που ακούσαμε από την Πολωνίδια Μεσελεβίτρια πριν από λίγο. Πάντω χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Οπότε από τη δικιά μα την πλευρά η αναφορά αυτή δεν μπορεί να κλείσει, διότι πρέπει να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Σε ένα πνεύμα βέβαια αμοιβαία κατανόηση και σεβασμού των αρμοδιοτήτων ε, και των δύο πλευρών, και τη Πολωνία δηλαδή και τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη δικιά μου την πλευρά αυτά είχα να πω. Α, συν ένα ότι η Πολωνία ρητά αναφέρει στο τέλος της απάντησής της ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε την ε, περίπτωση που από την αλλαγή αποφελωθούν κάποιοι πολίτες και μπορέσουν να συνάψουν ε, γάμο ή μόνιμη ένωση σε χώρα εκτός Πολωνίας, αυτές οι ενώσεις των πολιτών δεν θα αναγνωρίζονται στην Πολωνία. Οπότε δεν ερχόμαστε σε ένα άλλο πρόβλημα που είναι το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης τέτοιων συμφωνιών ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Uh, Μάλιστα. Προσφέρθηκαν οι διερμηνείς να κρατήσουν 10 παραπάνω λεπτά μαζί μας. Σας ευχαριστώ, κύριο Κάσμαν. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ το, την Πολωνίδα Διαμεσολαβήτρια Γι' αυτό που είπε πριν. Η διαδικασία εφαρμόζεται με διακριτικό τρόπο. Δεν έχουμε επιλύσει το πρόβλημα. Το θέμα της ομοφοβίας δεν ε, υπάρχει μόνο στην Πολωνία. Υπάρχει και σε κάποια από τα ιδρυτικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και απασχολεί τόσο πολύ την Κομισιόν και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό θέλω να σταματήσει. Λέω να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την ε, αναφορά. Χρειαζόμαστε ε, οι πολωνικές αρχές να επιλύσουν το πρόβλημα. Ευχαριστώ όμως και τη Διαμεσολαβήτρια και την, τους αναφέροντες που μίλησαν για αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να ανακατευτούμε στην νομοθεσία του κράτους μέλους, όπως το γαμικό δίκαιο. Είναι δική του αρμοδιότητα. Ο ρόλο μα είναι να ενθαρρύνουμε τι εξελίξει και να, σταματήσουμε, να σταματήσουν οι διακρίσει με τη δική μα βοήθεια και υποκίνηση. Ευχαριστώ και ευχαριστώ του αναφέροντε και τη διαμεσολαβήτρια και του διερμηνεί που μένουν παραπάνω. Και εγώ θα είμαι λοιπόν πολύ σύντομη. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά, να επιμείνουμε για το ποια είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Είναι το δικαίωμα τη ελεύθερη κυκλοφορία χωρί διακρίσει λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και αυτό συμπεριλαμβάνει ότι ο καθένας μπορεί όχι μόνο να κυκλοφορεί, αλλά ασκεί και τα δικαιώματά του καθώς μετακινείται. Γιατί αυτή η πρακτική είναι πρακτική διακρίσεων, θα πρέπει να σταματήσει. Όχι μόνο πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, αλλά πρέπει να στρεφόμαστε τακτικά προς την ε, Κομισιόν, ούτω ώστε να πηγαίνουν και αυτοί να συνομιλούν με τις πολωνικές αρχές για να υπάρχει μια κυκλοφορία, έτσι, μια κινητικότητα στο θέμα. Παρακαλώ. Σε αυτή την περίπτωση η διαμεσολαβήτρια έχει πάρει τη θέση. Μας εξήγησε ποια είναι η κατάσταση στην Πολωνία. Υπάρχει μια πρόοδος, μια κινητικότητα. Παραμένει ανοιχτή αναφορά. Απλώς ε, έχουμε πάρει κάποιες πληροφορίες και θα κρατήσουμε αυτές τις τρεις αναφορές μέχρι να λυθεί το θέμα. Ε, στην Πολωνίδια Μεσολαβήτρια, ευχαριστώντας και πάλι για την παρουσία της εδώ. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με την τελευταία αναφορά. Είμαι πεπισμένη ότι αυτή η αναφορά, αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί. Με βάση την ανάλυση μας, αντίθετα από την Κομισιόν, δεν πιστεύουμε ότι η νομοθεσία πρέπει να αλλάξει. Είναι θέμα πρακτικής περισσότερο, πρακτικής εφαρμογής και σωστών οδηγιών που πρέπει να δοθούν. Και θα πρέπει το Υπουργείο Εσωτερικών να εποπτεύει το έργο των αρμοδίων υπαλλήλων. Έχω παρενέβη και το Υπουργείο συμφώνησε ότι το πιστοποιητικό δεν είναι άδεια στο να προβεί κανείς σε γάμο η επίσημη συμβίωση. Και μετά από αυτές τις εξηγήσει πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες υποθέσεις και άλλες τέτοιες περιπτώσεις άρνησης έκδοσης αυτού του πιστοποιητικού. Εμείς ούτως ή έχουμε τακτές επαφές με τις οργανώσεις των ε, ομοφιλοφίλων ανδρών και γυναικών και των ε, φιλομεταβατικών. Αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις άρνησης, τότε θα έρθουμε σε επαφή με το Υπουργείο και θα δούμε αν η υπόσχεσή του ε, τηρήθηκε. Από νομική άποψη, νομίζω ότι το πράγμα είναι ξεκάθαρα. Απλώς πρέπει να δούμε τώρα τι θα γίνει στην πράξη. Ποιες θα είναι οι πρακτικές που θα ακολουθηθούν. Εγώ θα παρακολουθώ την κατάσταση. Αλλά κατά την άποψή μου, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουμε την νομοθεσία. Αυτό είναι το ένα λοιπόν. Το επόμενο. Είναι... Ευχαριστώ την κυρία Γκλέντς. Ξέρω την υπόθεσή της. Έχουμε παρέμβει τέσσερις φορές για αυτή την υπόθεση. Και μάλιστα πρόσφατα. Προσφύγαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε τέσσερις από τις πέντε υποθέσεις το Υπουργείο συμφώνησε μαζί μου. Πάντως έχουμε μια μόνιμη έτσι διαμάχη με το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Στις 30 ε, Αυγούστου φέτος έγραψε ένα γράμμα στον Υπουργό Εσωτερικών Θέλω να, θέσω, να παραθέσω δύο πράγματα από την επιστολή αυτή. Δεν θέλω να υποσκάψω το μηχανισμό επίδοσης των εγγράφων, ο οποίος ισχύει τώρα, ο οποίος εφαρμόζεται τώρα στην Πολωνία. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι ένδικα μέσα έχει στη διάθεσή του ο διάδικος. Θα πρέπει να δούμε όλες τις διαστάσεις ε, όλων των υποθέσεων, διοικητικών, αστικών και άλλων. Σήμερα οι πολίτες μετακινούνται πολύ περισσότερο από παλιά. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το κόστος επίδοσης των εγγράφων. Η πρώτη επίδοση θα πρέπει όμως να γίνει στο εξωτερικό. Και εν συνεχεία, ένας πληρεξούσιο στην Πολωνία θα πρέπει να προσδιοριστεί. Υπάρχουν όμως διάφορα νομικά προβλήματα, τα οποία ακόμα αντιμετωπίζουμε. Και με βάση τη νομική ανάλυση που κάνουμε, Θέλω να πω στην Επιτροπή σας ε, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ναι, όντως υπάρχουν προβλήματα. Μερικές φορές πρόκειται για νομικές παγίδες. Σε ορισμένε περιπτώσεις δεν υπάρχουν στη διάθεσή μας κάποιες ε, νομικές διατάξεις Φυσικά εμείς έχουμε κάποιες ιδέες για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Στις 19 Ιανουαρίου θα το συζητήσω με την πολωνική κυβέρνηση αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν διαφορές απόψεων. Εγώ έχω άλλες απόψεις από αυτές των Υπουργών. Ίσως και έρθει ο Πολωνός Επίτροπος από τη συνάντηση. Ε, μετά από αυτή τη συνάντηση μπορεί να καταφύγω, μπορεί να προσφύγω στο συνταγματικό μας δικαστήριο, ανάλογα με την έκβασή της. Γιατί είναι ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας μεταξύ της πολωνικής κυβέρνησης και εμού. Έχουμε και νομολογία, έχουμε κάνει και την νομική ανάλυση. Είμαι πεπισμένη ότι θα λυθεί τελικά αυτή η υπόθεση. Ίσως το νέο κοινοβούλιο την επιλύσει. Πολύ πιθανό όμως να προσφύγω και στο συνταγματικό δικαστήριο. Εξάλλου υπάρχει και η περίπτωση να αλλάξει ο, υπουργός, ε, ο νέος υπουργός... Ε, συγγνώμη, μπορεί να, αλλάξει πρακτική ο υπουργός ε, δικαιοσύνης. Καταλαβαίνει υπάρχει και το θέμα του κόστους Υπάρχει πραγματικά πρόβλημα, θα πρέπει να το επιλύσουμε. Αν σας ενδιαφέρουν όλες τις λεπτομέρειες, βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας. Σε ευχαριστώ όλους που παραμείνατε. Thank you,